Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, συνάδελφοι, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, περιμένουμε τον κύριο Παντσέρη, ο οποίος μόλις μπήκε στην αίθουσα. Buongiorno. Right. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Περνάμε στο πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης, έγκριση αυτής. Αφού δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνεται. Δεύτερον, ανακοινώσει του Προέδρου, δεν έχω κάτι να πω, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση. Και περνάμε στο τρίτο σημείο της μερικής διάταξης, σύσταση στο Συμβούλιο την Επιτροπή και την ΕΙΑΔ, ΕΙΕΔ σχετικά με τη Λιβύη. Ο συνάδελφός μας, ο κύριος Αντώνιο Παντσέρη, είναι η συγητής μας. 173 είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Έχει γίνει ήδη μια πρώτη συζήτηση μεταξύ του κύριου Παντσέρη και των Σκιωδών για να καταλήξουν σε 17 συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή να δώσω το λόγο στον κύριο ε, Παντσέρη για να μας πει που βρισκόμαστε στις συζητήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στο συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καταρχάς να ευχαριστήσω την γραμματεία της ΑΦΕΤ και του Σκιώδη για, το, θαυμάσια συνεργασία για ένα θέμα περίπλοκο όπως αυτό που από τη Λιβύη. Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, είχαμε διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην κατάθεση 17 συμβαστικών τροπολογιών που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των 173 173 τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Απλά και μόνο τώρα θα πρέπει να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης στη Λιβύη. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δείξουμε και να αναδείξουμε ένα ρεαλιστικό δρόμο λύσης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαπραγματεύσεις, όλες τις πρωτοβουλίες και όλες τις προσπάθειες που γίνονται. Βεβαίως υπάρχει και ταυτόχρονα το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών ως ε, μοναδική διέξοδος από την ορεινή κατάσταση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσουμε τη δυσκολία προσώπησης και τις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τωρινή κυβέρνηση Σεράρη Οπότε θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία μακρόπνοη κυβέρνηση εθνική συνένεση, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τι διαδικασίε ειρήνευση σε αυτή τη χώρα. Ταυτόχρονα τονίζουμε την ανάγκη και μάλιστα υποχρέωση, θα έλεγα, αναζήτηση ε, μια ευρεία προσπάθεια τι δικασιε ειρηνευση σε αυτη τη Λιβύη στα πλαίσια τη περιοχή Επίση τονίζουμε την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ζητώντα την υλοποίηση μιας μεγάλης διεθνούς διάσκεψης για τη Λιβύη, ταυτόχρονα αποτρέποντας τον μεμονωμένο πρωταγωνισμό κάποιων χωρών. Επίσης ζητάμε να γίνει ένας υποέλεγχο αφοπλισμός κάτι το οποίο αποτελεί την απαραίτητη προπόθεση για την επικοδόμηση οποιασδήποτε ειρηνευτική εθνική διαδικασία. Επίση, ενθαρρύνουμε έντονα τη διοργάνωση εντό του 2018 με ε, διεθνή ε, μια διεθνή ε, διάσκεψη μέσα στο 2018 με την βοήθεια τη Επιτροπή Βενετία και με διεθνή υποστήριξη ώστε να καταλήξουμε ακριβώ αυτό το πλαίσιο σταθερότητα τη χώρα. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε την σημασία τη ταχεία έναρξη μια όσο πιο ευρεία διαδικασία γίνεται που θα περιλαμβάνει όλε τι φυλέ και τι τοπικέ οργανώσει, ώστε να οικοδομηθεί επιτέλου μια ελεύθερη και δημοκρατική Λιβύη. Καταδικάζουμε επίση τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων στη χώρα. Ταυτόχρονα δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μα όσον αφορά την θητεία και την εντολή του Διεθνούς Οικαστηρίου. Τώρα για την μετανάστευση και το θέμα της εσωτερικής μετανάστευσης και των προσφύγων θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ροές από και προς τη χώρα. Και τέλος, υπό το φως αυτών προσπάθησα να σας ε, περιγράψω νωρίτερα, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει και σήμερα βεβαίως θα ακούσουμε προσοχή τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις των σκηνοδών εισηγητών και των υπολείπων συναδέλφων που θα ήθελα να παρανεύουν, με την ευχή βεβαίω η έκθεση αυτή να πετύχει τη μέγιστη τη συνένεση και σύγκληση ξεκινώντας από την ψηφοφορία αύριο το πρωί στην Επιτροπή μα. Αυτά προεδρεπομένα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, uh, Ευχαριστούμε. We have an indicative duration. 10 λεπτά είναι η ενδεικτική διάρκεια που έχει προβλεφθεί για αυτό το σημείο. Και έχω αυτή τη στιγμή πέντε συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο Στετίνα, Τένακ, Λόχμπίλαρ, Κόσο και Καστάλτο. So we have Mr. Bettini Ο κ. και ο κ. Χατζηγεωργίου επίσης. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Όχι. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε τελειώσει από και 10. Είναι ήδη και 20 και έχουμε 7 ομιλητές. Δύο λεπτά στον καθένα. Δύο λεπτά στον κάθε ομιλητή. Κύριο Στετίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Καταρχήν ευχαριστήσω τον κύριο Παντζέρη και τους άλλους συναδέλφους από τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες που έλαβαν μέρος. Ε, ασχολούμαι τη Λιβύδο και αρκετό καιρό και έχουμε μάλιστα γνωρίσει και ένα συνέδριο σχετικά με την κατάσταση στη χώρα αυτή. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιε είναι οι ανάγκες, προκειμένου να βοηθήσουμε τη χώρα να εξασφαλίσει σταθερότητα και ασφάλεια των πολιτών της και την ασφάλεια των ε, προσφύγων και μεταναστών. Μέχρι τώρα οι σκιώσεις ηγητές συναντήθηκαν μία φορά μόνο και στο πλαίσιο της διαδικασίας συμβιβασμού συμφωνήσαμε ως ΕΛΚ στις ε, επί των προτάσεων ε, που έγιναν. Ε, Δυστυχώ δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε την, ε, τον κατάλογο ψηφοφορία. Θα θέλαμε να ζητήσουμε να αναβληθεί η ψηφοφορία, αλλά έχουμε, βρει, έχουμε συμφωνήσει. Θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τους συναδέλφους. Καλή επιτυχία στην, ε, συνεδρία, στην ψηφοφορία αύριο. Ο κ. Στάνοκ έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομο Και εγώ ήμουν στη συνάντηση των σκιωδών συγητών που συζητήσαμε τις συμβαστικέ τροπολογίες. Ε, είμαι μία από, τις, ε, από μία από τις δύο βασικές χώρες που παρενέβησαν στρατιωτικά στη Λιβύη. Δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της εξωτερικής πολιτικής της Βρετανίας ή της Γαλλίας η Λιβύη αποσταθεροποιήθηκε από τότε ε, πλησιάζει στο να είναι ένα κατεστραμμένο και αποτυχημένο κράτος στην πολιτική μου ομάδα το συζητήσαμε μακρόν το θέμα ε, με διαφορετική άποψη από τους φιλελεύθερους εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το πρόγραμμα δράσης του ΟΗ για τη Λιβύη και την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας καθώς επίσης και το ρόλο του κ. Σαλάμι, του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ. Η Λιβύη εξακολουθεί να είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι αρκετά κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα λαθρεμπορίου, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, τζιχαντισμό, ε, τρομοκρατία, ο Ισλαμικός στρατός έχει στήσει γερά τα πόδια του στη και το Ιράκ. Σημαντικά προβλήματα λοιπόν σε σχέση με την σταθεροποίηση της χώρας Υπάρχει και ε, ένα ταμείο επίγουσα βοήθεια ε, ε, για τη Λιβύη και το αντίστοιχο του ΟΕΕ. Εθνών. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για να, βρούμε, να, ξα, ζητήσουμε μια σταθερότητα και να επιστρέψουμε στο κράτο δικαίου και τη δημοκρατία. Μακροπρόθεσμα βέβαια εντωμεταξύ. Α διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί τουλάχιστον να λειτουργεί με ασφάλεια παρέχοντα ανθρωπιστική βοήθεια ε, με επανεγκατάσταση ε, των ε, μετακινούμενων πληθυσμών προκειμένου να καταπολεμήσουμε την διεθνή τρομοκρατία κλπ. Η έκθεση είναι ισορροπημένη και στηρίζουμε τις, τους συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. The Green Group... Η πράσινη είναι πιο πολύ από την ΚΟΕ αυτή τη στιγμή. Είναι πιο πολύ από την ΚΟΕ πλέον, οπότε ε, Κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε και τον συγχωρητή τον κύριο Παντσέρη που ηγείται της διαπραγμάτευσης και τον ευχαριστούμε που ενσωμάτωσε πολλές από τις τροπολογίες της ομάδας μας στις συμβαστικές τροπολογίες. Ιδίως τις προτάσεις μας που επικεντρώνονται στο ρόλο των γυναικών και των μειονοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί μια σταθερή μακρόπνοη πολιτική συμφωνία και την προειδοποίησή μας προς τους ε, περιφερειακούς παίκτες να μην ε, επιδίδονται σε στρατοτική δράση χωρίς ε, συνεννόηση. Επίσης, καλούμε την Λιβύη να υπογράψει την Σύμβαση της Γενέβης του 1951 για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να υποστηρίξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά ε, βεβαίως στο στο πλαίσιο των συμβασμών. δυστυχώ όμως δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις συμβασικές τροπολογίε που αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση στη Λιβύη. Για παράδειγμα, εμείς δεν μπορούμε να ε, ε, υποστηρίξουμε την έκκληση που γίνεται για ενίσχυση της συνεργασίας ΝΑΤΟ και ε, της επιχείρησης Σοφία. Ε, επίσης δεν υποστηρίζουμε τις αποστολές κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και δεν υποστηρίζουμε την, ε, την ενίσχυση της ε, λιβικής ε, ακτοφυλακής που εμπεριέχεται στο κείμενο. Παρ' όλα αυτά προσβλέπουμε στο, στο να ψηφιστεί η έκθεση αυτή και ελπίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Παντσέρη, διάβασα μόλις πληροφορίες ότι ε, ο Χαφτά της Λιβύης είναι βαριά άρρωστος. Αυτά μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και, για, τον πολιτικό κόσμο και για το στρατιωτικό κόσμο της Λιβύης. Αυτά σας παρακαλώ να τα πάρετε υπόψη σας γιατί μπορεί να καταστεί παροχημένο το κείμενο στο οποίο θα καταλήξουμε. Ευχαριστώ. Σκιώδης για την ΚΟΕ είναι ο κύριος Κούζο. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Είπαμε στον κύριο Παντσέρη ότι περιέχει θετικά και λιγότερα θετικά στοιχεία η δουλειά του. Τώρα βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες του κοινοβουλίου να ζητούν να παλευθεί στη Συρία αυτό που γίνει στην Λιβύη. Η ε, Λιβύη που έχω μια αποτυχημένη χώρα, ε, μεγάλη έλλειψη σταθερότητα στην χώρα, ε, χώρα εξαφανισμένη, χώρα κατακαιρματισμένη, με φυλές, με σκλαβοπάζαρα και μάλιστα αυτή τη στιγμή οργανώνεται και η δημιουργία του Ισλαμικού κράτους, ΔΑΕΣ. Στην Ολομέλεια θα έπρεπε να έχουμε μια ευρεία συζήτηση για αυτά τα θέματα, πάντως εμείς θα υποστηρίξουμε κάποιες από τις τροπολογίες της σύστασης, αλλά ξεκάθαρα βέβαια είμαστε κατά κάποιων άλλων ε, στοιχείων που αφορούν τη Λιβύη και ιδιαίτερα αυτή η δύναμη η συνοριακή που όπως μας έλεγαν οι ΜΚΟ τις, τις περασμένες εβδομάδες που διασώζουν τους ε, πρόσφυγες μετά από την εξάστρωση της επιχείρησης Μαρενόστρομ αυτό ε, που συμβαίνει είναι ότι αναθέτουν την ε, απόθεσή τους σε εγκληματίες που τους πυροβολούν για να μην πάνε στην Ευρώπη. Είναι πειρατές αυτοί, τους οποίους εξοπλίζουν και με αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και γι' αυτό και στο λόγο στα συγκεκριμένα σημεία θα απέχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Καστάλντο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Παντσέρη για θαυμάσια δουλειά του και το καλό αποτέλεσμα που πέτυχε παρά τις αποκλίσεις στις απόψεις μεταξύ των διαφόρων σχεδόν εισηγητών. Πέρα από τις προτάσεις και τις συστάσεις, όπως λέγαμε προηγουμένως τους συναδελφούς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την είδηση για το θάνατο του στρατηγού Αφτάρ, ε, που μετά διαψεύστηκε. Κάτι το οποίο όμως βέβαια συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση της χώρας και στην αύξηση της μεσαγειακής κρίσης. Νομίζω ότι αυτό οδηγεί σε νέα σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν την ευαίσθητη ισορροπία στη Λιβύη. Γιατί η ενδεχόμενη εξαφάνιση του ή θάνατό του θα μπορούσε βεβαίω να διαταράξει την τωρινή κατάσταση των πραγματεύσεων. Εξάλλου υπάρχει και υψηλό κίνδυνο κατακαιρματισμού όσον αφορά την ε, πάλι για την εξουσία στο εσωτερικό αυτών των ομάδων που αφορά τους, τον κύκλο του στρατηγού Αφτάρ, που πάλι αυτή δεν αφορά μόνο βεβαίω την διαδοχή, αλλά κυρίω του φυσικού πόρου τη χώρα, το πετρέλαιο δηλαδή. Θα πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη μα το γεγονό ότι η νέα χαόδη ε, κατάσταση ε, θα οδηγήσει στην ε, επαναφορά νέων δυνάμεων, οι οποίε δεν έχουν ακόμα αιτηθεί και το οποίο θα αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώ οι συζητήσει που θα έχουμε στην Ολομέλεια θα πρέπει να λάβουν υπόψη του τα στοιχεία αυτά και θα πρέπει να ενημερωθεί κατά κάποιο τρόπο η έκθεση όσον αφορά το προσδοκόμενο πλαίσιο που θα αλλάξει τις επόμενες μέρες. Εγώ δεν μπορώ παρά να στηρίξω και να συμφωνήσω με το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών, το μόνο εφαρμόσιμο δηλαδή για την σταθεροποίηση της χώρας και την έναρξη της διαδικασίας ειρήνευση στην χώρα μας με τον αφοπλισμό των παραστατευτικών ομάδων. Επίσης, έχουμε και διάφορες χώρες οι οποίες μέχρι τώρα δεν βοήθησαν να βρούμε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τους Γιώδης. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές. Ο κύριος Μπετίνη, ο κύριος ε, Χατζηγεωργίου και ο κύριος Σάφχαουζα. Ευχαριστώ. Πρώτον, κλείνω τον κατάλογο ομιλητών. Κύριε Μπετίνη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Να πω μόνο ότι η έκθεση αυτή μου φαίνεται πολύ καλή, συγκεκριμένη και νομίζω αποδεικνύει μια γνώση της κατάστασης, όχι μόνο στη Λιβύη, η οποία είναι νομίζω σημαντική. Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξει μια ισχυρή σύγκληση, ώστε εμείς να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε μια κατάσταση πλήρου σύγχυσης, ώστε να δείξουμε ότι έχουμε ομόνια, ότι ομονοούμε μεταξύ μας όσο γίνεται βέβαια. Εγώ να τονίσω μόνο ότι αυτές οι συστάσεις μας θα πρέπει στη συνέχεια βεβαίως να συνδυαστούν με τις πρωτοβουλίες και την βούληση αυτών που κάνει αυτή τη στιγμή η Ιταλία και που θα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες επειδή η Ιταλία είναι η χώρα η οποία εμπλέκεται αμεσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση αυτή λόγω ακριβώς των ιστορικών και γεωγραφικών σχέσεων που έχει η χώρα αυτή τη Λιβύη. Ευχαριστούμε κύριε Μπετίνη. Ο κύριος Χατζηγεωργίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντζέρη για την έκθεσή του η οποία πράγματι έχει αρκετά θετικά στοιχεία, μερικά τα οποία κρίνουμε αρνητικά θα δούμε αύριο πώς ε, ψηφίζουμε σε αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα κι εγώ από όσα έχουν λεχθεί για το χάος που επικρατεί στη Λιβύη, οργανωμένο έγκλημα, κυρίως επιστροφή του τζιχατισμού, σκλαβοπάζαρα, διαφθορά, τρομοκρατία. Ένα απίστευτο χάος και σε όλα αυτά ο πιθανός θάνατος του Αφτάρ νομίζω και εγώ ότι θα συμβάλλει αρνητικά στις ε, εξελίξεις στην περιοχή. Ήταν ένας άνθρωπος στρατιωτικός που επηρέαζε κατά τις ε, εκθέσεις του Κοινοβουλίου θετικά την κατάσταση. Έχω μόνο μία ερώτηση. Αυτές οι συστάσεις που περιέχει η έκθεσή μας και που θα ψηφιστούν, πώς θα εφαρμοστούν, τι πιστεύουμε γι' αυτό, ποια στοιχεία έχουμε ότι θα υλοποιηθεί μέρος τους. Αυτό είναι το το σημαντικό κομμάτι. Και κλείνω λέγοντας ότι δεν θα κάνω αναφορά στις ευθύνες που υπάρχουν σε κράτη-μέλη για το τι επικρατεί σήμερα στη Συρία. Και θα έπρεπε ε, μερικοί εκπρόσωποι αυτών των κρατών μελών να μας έλεγαν, να, να, να κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ταχύτατα. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη, είναι πολύ εύκολο να αποσταθροποιηθεί μια χώρα και πολύ πιο δύσκολο να ανοικοδομηθεί. Αυτό που κάναμε στη Λιβύη φαίνεται αδύνατο σήμερα, δεδομένου το ότι δεν υπάρχουν πια ηγέτες. Φανταστείτε λοιπόν την ίδια κατάσταση στην Συρία αν φύγει ο Ασάντ θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση και θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στην ανοικοδόμηση της χώρας, γιατί θα λείπουν ακριβώς τα βασικά στοιχεία της ανοικοδόμησης. Δεύτερη παρατήρηση, χωρίς κράτους είναι απολύτως αδύνατο να δοθεί βοήθεια για την ανάπτυξη. Δεν, δεν μιλάμε για τις ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Και θα μπορούσα να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη αναποτελεσματικότητα στην διαχείριση της βοήθειας αυτής όσον αφορά κοινωνία πολιτών και πληθυσμό. Τρίτη παρατήρηση. Με το θάνατο του στρατηγού Αφτάρ, στο ενδεχόμενο αυτό έτσι, δεν ξέρω ακριβώ πώς έχει η κατάσταση, παρόλο που έχω επαφές με, τους, με το προσωπικό του, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, αν ισχύει αυτό, μου φαίνεται τελείω αδύνατο να πετύχουμε την ανοικοδόμηση. Είμαι πολύ απεσιόδοξο, γιατί είχαμε ένα στρατηγό στον οποίο μπορούσαμε να βασιστούμε. Έτσι, ανεξάρτητα με το τι λέει η έκθεση, αυτέ οι σχέσει θα μα επέτρεπαν να ανοικοδομήσουμε την χώρα. Και αυτό το βασικό στοιχείο θα λείπει πια. Και φοβάμαι ότι η αποσταθεροποίηση που επέβαλε η Δύση σε αυτή τη χώρα να είναι απαγορευτική και δεν θα υπάρχει λύση δυστυχώς. Σας ευχαριστώ. Okay, thank you, Mr. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Παντσέρη, θέλετε να απαντήσετε όσο γίνεται πιο σύντομα, παρακαλώ. Ταχύτατα, ναι. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συμβολή και τη διαθέσή τους. Δύο διευκρινήσεις μόνο. Εγώ από ό,τι ξέρω, ο Χαφτάρ δεν έχει αποβιώσει. Έκανε μια εγχείρηση καρκίνου και είχε και μια πλευρίτιδα η οποία επιβάλλει την υγεία του. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παραμένει στην λιβική πολιτική σκηνή. Βεβαίω, αν τύχει τώρα κάτι το ιδιαίτερα αρνητικό, συμφωνώ με του υπόλοιπου ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε κάπω αυτή την έκθεση, γιατί η κατάσταση βεβαίω αλλάζει ριζικά. Και τέλο, πώ θα μπορούσαμε να κάνουμε απαιτητή αυτή την σύσταση, δηλαδή ώστε να τη προσδώσουμε μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο Κοινοβούλιο και να δεσμεύσουμε το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν ώστε η σύσταση αυτή να ακολουθηθεί στα πλαίσια τη εξωτερική πολιτική. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε, σε αυτό πρέπει να στοχεύουμε. Ευχαριστώ πολύ παντό, ευχαριστώ όλου σα. Okay. Ωραία. Σα ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σύντομη συζήτηση. Η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα γίνει αύριο το πρωί. Και στην Ολομέλεια θα γίνει στην, την εβδομάδα 11 με 14 Ιουνίου. Πολύ ωραία και περνάμε στο επόμενο σημείο. Σημείο υπαριθμών 4. Σύσταση στο Συμβούλιο σχετικά με την Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής που βρίσκεται υπό διαδικασία εξυγχρονισμού. 69 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Η ε, είναι ο κύριος Τσάρλ Τάνοκ, 25 είναι οι συμβαστικές τοπολογίες που προτείνει. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά που ανέλαβα αυτή την έκθεση. Η Χιλή είναι ε, χώρα την οποία επισκέφθηκα πριν από πολλά χρόνια σε πιο σκοτεινές εποχές και έκτοτε την έχω παρακολουθήσει να ανθίζει ε, ως δημοκρατία και ως οικονομία στη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό και με μεγάλη μου χαρά ανέλαβα το καθήκον της ε, σύνταξης αυτής της έκθεσης για, για τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής. Είμαι τόσα χρόνια εδώ που θυμάμαι και την πρώτη τέτοια συμφωνία σύνδεσης που είχε ε, υπογραφεί πριν από 20 χρόνια. Ο κ. Αλαφράνκα τότε ήταν εισηγητής. Βλέπουμε πλέον ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες και με το Μεξικό και με τη Χιλή ε, και η ΑΦΕΤ ασχολείται με όλα τα ζητήματα διαλόγου και συνεργασίας με τη χώρα αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τους Σκιώδης. Ξέρω ότι είναι μικρό, πέντε είναι μόλις οι συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό όμως αντικατοπτρίζει και τον γενικά ε, συνολικά μικρό αριθμό τροπολογιών που κατατέθηκαν, 69. Ε, και εγώ 16 ε, ε, δέχομαι από αυτές τις τροπολογίες από τις 38 ε, που δεν κατέστη δυνατόν να ενσωματωθούν στις συμβαστικές τροπολογίες τις υπόλοιπες δεν τις δέχομαι για διάφορους λόγους αρχικά είχα σκοπό να υπερψηφίσω την τροπολογία των πρασίνων υπαριθμών 19 στη συνέχεια όμως συνειδητοποίησα ότι τεχνικά και από άποψη πραγματικότητας δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο γιατί η ΕΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Χιλη. Ε, και με αυξανόμενο βεβαίως το ρόλο της Κίνας που έχει διεισδύσει όπως στην Λατινική Αμερική και με τη Βραζιλία συμβαίνει το ίδιο. Δεν ξέρω αν οι πράσινοι ε, θέλουν να αποσύρουν την τροπολογία τους ή εν πάση περιπτώσει με προφορική τροπολογία να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κατάλληλη ε, τροπολογία προφορική. Είπα ότι βασίζομαι στο γεγονός ότι η Χιλή είναι μια προηγμένη δημοκρατία και αποτελεί σοβαρό πολιτικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Γι' αυτό και ελπίζουμε όλοι να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι όσο, πιο γίνεται, όσο γίνεται πιο θετικό, θα αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που έχουν γίνει στη χώρα ε, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Από την επιστροφή, την αποκατάσταση της δημοκρατίας έπειτα από την πτώση της ε, στρατιωτικής δικτατορίας υπό τον στρατηγό Πινοσέτ. Εκεί όπου οι τροπολογίες ε, ήταν υπερβολικά περιγραφικές και εξέφευγαν από το πεδίο της ε, έκθεσης ή θεωρώ ότι είναι πολύ αρνητικές, δεν τις υποστηρίζω. Παρ' όλα αυτά περιμένω να ακούσω τα σχόλια των ε, συναδέλφων και, και των σκιωδών για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περιττέρω την έκθεση αυτή και όπως είπαμε η ψηφοφορία είναι αύριο. Ευχαριστώ Τσαρλ Στάνοκ Περνάμε τώρα στους ομιλητές. Έχουν ζητήσει το λόγο η κυρία Ζόφκο και ο κύριος Καστάλτο. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Όχι. Περνάμε λοιπόν στον ε, σκιώδη του ΕΛΚ, την κυρία Ζόφκο. Ευχαριστώ πολύ έχοντας υπόψη τη σημασία του εξοχρονισμού της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής με καλύτερες βελτιωμένες ε, διατάξεις εμπορικής και ε, τομεακής συνεργασίας αλλά και συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας θεωρούμε ότι αυτή, αυτός ο εξοχρονισμός μπορεί να αναβαθμίσει την συμφωνία. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες χαιρετίζουμε τις συμβαστικές που έχει προτείνει ο κ τον Τάνοκ θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένες και έλαβαν υπόψη τις θέσεις του ΕΛΚ στα πιο σημαντικά ζητήματα. Επιπλέον, λόγω και της επίσκεψής μου στη Χιλή, στις αρχές του χρόνου, ε, εγώ ε, έχω συναντηθεί με σημαντικό αριθμό ε, μελών της, της χιλιανής παρικίας σε όλο τον κόσμο και ε, υποστηρίζουμε ιδίως ε, τις αναφορές της έκθεσης ε, στην έρευνα, τον πολιτισμό, την παιδεία και όπως σημειώνει, σημείωσε μάλλον ο εισηγητής, βλέπουμε ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη Χιλή προκειμένου να διατηρήσουμε έστω σε έναν βαθμό την επιρροή μας στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζόφκο, κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω τον συγητή Τσάλ Στάνοκ για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε στην έκθεση αυτή. Σήμερα οι συμφωνίε σύνδεση με Χιλή, όπω και αυτή με το Μεξικό, είναι ιδιαίτερα σημαντικέ, ενισχύουν τον ρόλο τη Ευρώπη ω εταίρου κλειδί στη Λατινική Αμερική, τη στιγμή που η παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο αβέβαιη και άλλε χώρε έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή, όπω η Κίνα, που όπω ακούσαμε είναι ο πρώτο εμπορικό εταίρο τη Χιλή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή ανανέωση τη φιλία μα με τη Χιλή, με τη Χιλή όπω και για να αντιμετωπίσουμε διάφορε παγκόσμιε προκλήσει, μετανάστευση, περιβάλλον κλπ. Επίση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογό μα που έχουμε ξεκινήσει με το 2009 με αυτή τη χώρα και προτείνω που και χαίρομαι που τροπολογίε που κατέθεσα όπω 28 είναι αποδεκτές, ιδιαίτερα αυτοί που ρυθμίζει το θέμα των Μαπούτσε, που στη γλώσσα του σημαίνει λαός της γης. Είναι μια φυλή που επιβίωσε της ευρωπαϊκής απίκησης. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να χάνουν, να τους αφαιρούν, να τους αποσπούν εδάφη και τα εδάφη τους συνεχίζονται να καταλαμβάνονται από την κυβέρνηση και τους στρατούς Χιλής για να δημιουργηθούν ε, χώροι βοσκής. Στην 31 επίσης τονίζω την ανάγκη ενθάρρυνσης της χελής για την έναρξη μιας σωστής διαδικασία που θα αντιμετωπίζει τα θέματα της τρομοκρατίας. Έχουμε ακόμα ε, ορισμούς στην νομοθεσία που προέρχονται από την εποχή του Πινοσέ ε, με ευρείες ε, έννοιες και ορισμούς και, που επιτρέπουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως κατά των φυλών που ανέφερα προηγουμένως. Είχαμε μάλιστα και συλλήψεις ε, ε, ηγετών ή εκπροσώπων των Μαπούτσι που αναγκάν να μετακινούνται συνεχώς. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση τη Χιλής να αναθεωρήσει την νομοθεσία αυτή, ώστε εκτός από τη γη να μην χάσουν και την ελευθερία τους αυτοί οι φίλοι Μαπούτσι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Θα το λόγο. Όχι. Τζον Στάνοκ, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ τους δύο σκιώδης ηγητές ε, για τα ενθαρρυντικά του σχόλια. Στον συνάδελφο από το ΕΛΚ έχω, ήρθα σε επαφή με την ε, ε, διασπορά, κροατική διασπορά στην Χιλή που είναι μάλιστα και ιδιαίτερα πετυχημένη επιχειρηματικά. δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε αυτές, αυτούς τους δεσμούς σε όλη τη Λατινική Αμερική υπάρχουν μεγάλες κοινότητες ε, ε, ατόμων που κατάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι άνθρωποι που έχουν δεσμούς με την Ευρώπη, δημιουργούν τουρισμό κλπ. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο κ. Καστάλντο, ε, σημείωσα τα όσα είπε για τους αυτόχθονες, τους Μαπούτσε, τους προκολομβιανούς ε, κατοίκους της ε, ε, Λατινικής Αμερικής κλπ. Είναι πολύ σωστό που αναφέρει πως πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Η Συμβαστική Τροπολογία Υπαριθμών 1 αυτό ακριβώς έχει ως στόχο να μπει στην έκθεση ένα τέτοιο σχόλιο. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι άλλο και ελπίζω ότι αύριο το κείμενο θα ψηφιστεί με πολύ ευρεία πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Πράγματι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί, παρόλο ότι στην Ολομέλεια θα γίνει η ψηφοφορία τον Ιούνιο. Περνάμε στο σημείο 5. Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή εκλογικών παρατηρητών για την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών τη 15η Απριλίου στο Μαυροβούνιο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καστάλντο που ήταν επικεφαλή, να σα υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο συζητήσαμε με τον Ζόραν Παζίν τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Δικαιοσύνης του Μαυροβουνίου εδώ σε αυτήν την Επιτροπή. Είχαμε συζητήσει για την ε, σημασία των προεδρικών εκλογών που θα είχαν ως στόχο την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα. Κύριε Καστάλτο, αναφέρετε μας για την εμπειρία σας και μετά θα ακούσουμε και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, χαίρομαι που σας κάνω αυτή την ενημέρωση ακριβώς τη μέρα που συζητιέται στην Κομισιόν εκ μέρους του Επιτρόπου το πακέτο για τη διεύρυνση. Αυτή λοιπόν η ενδεχόμενη αποστολή παρατηρητών Επιβεβαιώνεται ότι είναι απαραίτητο και για τα Βαλκάνια και ε, για την Όση να υπάρχει κάτι τέτοιο Τέλος, στο τέλο ο κ. Τσουκάνοβη βέβαια με το, στον πρώτο γύρο και στι εκλογέ με 53,9%. Πρέπει να σα πω ότι αυτέ οι εκλογέ ήταν υψηλού επίπεδου, κατά τη διάρκεια των οποίων τα βασικά δικαιώματα και οι διεθνεί προδιαγραφέ υπερτηρήθηκαν, λέει ο Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Από τη στιγμή που είχαμε μια μακρά περίοδο ε, αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων του 2016 και μποϊκοτάζα τη Είχαμε μάλιστα και διαχείριση αυτών των εκλογών που ήταν στο ύψος των περισσότερων χώρων της Ένωσης. Έγιναν λοιπόν με ηρεμία αυτές οι εκλογές και είχαμε πάει σε τρία μέρη. Στην Ποτκόριτσα, στις ακτές και στο εσωτερικό της χώρας, στο Κόλασαν και στον Περάνε. Οι ομάδες ε, παρατηρητών λοιπόν αποτίμησαν θετικά το μέγιστο μέρο των διαδικασιών με ελάχιστε παρατυπίε που, ε, που είναι βέβαια δεν επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Και η μόνη παρατήρηση που είχαμε ω αποστολή αφορούσε τι κάλπε, οι οποίε κάλπε τι θεωρήσαμε όχι ασφαλεί και ιδιαίτερα ευάλωτε, εύθραυστε. Οπότε εύκολο, εύκολα θα μπορούσε κανεί να ρίξει μέσα παράνομα ε, ψηφοδέλτια στις κάλπες αυτές αλλά θεωρούμε τέλο πάντων σε αυτό το σημείο όσον αφορά την σύνθεση των υλικών που αποτελούν τις κάλπες θα μπορούσε να βελτιωθεί. Και ο πρώτο μάλιστα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερε αρμοδιότητες στο σύστημα του Μοντενέγκρο και πέτυχαν να κάνουν εκλογές χωρίς εντάσεις και μάλιστα η προεκλογική περίοδο ήταν πολύ σύντομη. Είχαμε και κατάθεση των ψηφοδελτίων σχετικά καθυστερημένα. Έχουμε και τις τοπικές εκλογές ε, στις 27 του Μάη που θα καλύψουν το 70% του εκλογικού σώματος, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Παγκόσμια, που θα αποτελούσαν άλλο ένα πολιτικό τεστ. Ήταν λοιπόν υποδειγματικές οι εκλογές. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι και ο κύριος ε, Τσοκάνοβιτς ε, είχε και, μια, είχε και ένα σημαντικό θεσμικό πλεονέκτημα. Όπως μας είπαν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, έχουν την εντύπωση ότι οι υποψήφοι της πλειοψηφίας έχουν κάποια πλεονεκτήματα παραπάνω λόγω ακριβώς της ε, αλληλοσύνδεσης μεταξύ κυβέρνησης και διοίκησης σε σχέση με τους υπολείπους ε, υποψηφίους που καμιά φορά παρουσιάζουν και αυτό το θέμα καμιά φορά οδηγεί σε ελαδιακές σχέσεις. Είχαμε και τι συστάσει του ΟΝΤΙΡ και τη Επιτροπή τη Βενετία. Κάποιε από τι συστάσει του 16 του 17 έγιναν δεκτέ από το Κοινοβούλιο του Μοντενέγκρο, αποδεικνύοντα μια αντίστοιχη πολιτική βούληση. Όμω κάποιε συστάσει δεν ήταν δυνατόν να γίνουν αποδεκτέ λόγω ακριβώ του μποϊκοτά τη αντιπολίτευση που δεν επέτρεψε στο Κοινοβούλιο να διαθέσει το, απαραίτητα δύο τρίτα για την υλοποίηση κάποιων αλλαγών. Θεωρούμε λοιπόν ότι κάποιες αλλαγέ μικρέ θα έπρεπε να είχαν γίνει, όπως αυτό που ανέφερε προηγουμένως για τις κάλπες, επίσης το θέμα της εθνική Εκλογικής ε, Επιτροπής και αυτό συνδέεται και με το δεύτερο σημείο που θα θέλω να θίξω, δηλαδή η επαγγελματικότητα και διαφάνεια κάποιων κρατικών οργάνων όπως η Εθνική Εκλογική Επιτροπή και η Αρχή για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα εκεί μας απαγοήτευσαν και η εργασία της ε, Εκλογικής Επιτροπής ε, πολλές φορές δεν ήταν διαφανής. Ε, πρέπει όμως να είμαστε βέβαιοι σε αυτά που λέμε, επειδή ακριβώς γινόταν και κλεισμένο το θηρόν συναντήσεις και πρακτικά δεν δημοσιεύονταν. Και επίσης ενημερωθήκαμε στη συνέχεια ότι για την αθέτηση μέτρων διαφάνειας δεν είναι απαραίτητη η παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Οπότε στην ουσία οι, οι της εκλογικής επιτροπής μας είπαν ψέματα. Επίσης, αντίστοιχα, δεν απάντησαν πιστικά οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Καταπολέμησης ε, της Διαφθοράς. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση κάποιων ε, υποψηφίων, ιδιαίτερα όταν εμεί καταδείξαμε κάποιες ελλείψεις σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Επίσης, ο Πρωθυπουργό Μάρκοβιτς έχει κάποιο συγγενή σε αυτή την επιτροπή που ανέφερα προηγουμένω. Και δεν μπορούσαμε εμεί ω ε, παρατηρητέ βεβαίω για αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα. Ε, θα πρέπει, ξαναλέω, να, υπάρχουν, να υπάρχει επαρκή χρόνο για τι εκλογικέ διαδικασίε, για την ε, προεκλογική περίοδο και την προβολή των υποψηφίων. Ο κύριος εκπρόσωπος της ε, αντιπολίτευσης διέθεσε μόνο το 1 τρίτο του χρόνου του και ο κύριος ε, Τζουκάνοβιτ δεν συμμετείχε σε όλες τις εκπομπές που προβλεπόταν. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί βεβαίω την ε, διαφάνεια. Επίσης να πω κάτι για τα οπτικοακουστικά. Το Κοινοβούλιο αντικατέστησε δύο μέλη του αντίστοιχου Εθνικού Ραδιοτηλεπτικού Συμβουλίου λόγω σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι το οποίο βεβαίως αποτελούσε και μια πρόκληση για την αυτονομία αυτών των οργάνων στα πλαίσια μιας προσπάθειας πολιτικοποίησης αυτών των οργάνων. Και τέλος να πω δύο λόγια για τους υποψηφίους. Συναντήσαμε 7 υποψηφίους, μεταξύ των οποίων ε, μια κυρία, μια γυναίκα, την κυρία Βουξάνοβιτς, που παρόλο που προερχόταν από την αντιπολίτευση, κατάφερε να φτάσει στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι οι παρόντες συνάδελφοι μπορούν ακριβώς να επιβεβαιώσουν αυτά που νιώσαμε όλοι σε αυτή την ε, συνάντηση, ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι της ε, αντιπολίτευσης είχαν στόχο βεβαίω ε, την ήττα της κυβέρνησης, χωρίς όμως να έχουν ένα πιστικό, εναλλακτικό πολιτικό πρόγραμμα. Ήταν υπέρ του ΝΑΤΟ επίσης και κατά της Ρωσίας και της Σερβίας. Είδαμε επίσης κατά των επαφών μας, μιλώντας με τον κόσμο, τους πολίτες, ότι υπάρχει μια μεγάλη ε, τάση, μια μεγάλη έφεση προς την Ευρώπη. Μεγάλο ποσοστό των πολιτών της χώρας θέλουν να γίνουν μέλος της Ένωσης και έχουν μια πολύ θετική στάση. Και θεωρούμε ότι είναι προς κάθε συμφέρον της Ένωσης να ικανοποιηθεί, να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα και ακριβώς θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό προς τον κύριο Τζουκάνοβη, τον πρόεδρο, σε μία από τις επερχόμενες ολομέλειες. Ευχαριστώ. Uh, Με ταχύτητα ρεκόρ μιλήσατε κύριε Καστάλτο. Ευχαριστούμε. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο, κύριο κύριος Πίτουλα, κύριος Τάνοκ. Κανείς άλλος, αυτοί οι δύο. Παρακαλώ κύριε Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Καστάλντο όσον αφορά τις προεδρικές ε, εκλογές στο Μαυροβούνιο. Εμείς οι 7 ε, ήμασταν ε, μεταξύ των 2.000 ξένων παρατηρητών που ήλεγξαν τις ε, εκλογές στο Μαυροβούνιο από διεθνείς οργανισμούς. Είναι οι πρώτες μεγάλες εκλογές μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές που έγιναν το 2016 ε, που πραγματοποιήθηκαν υποδραματικές ε, περιστάσεις και φαίνεται ότι αυτές, αυτή η εκλογική μάχη κύλησε πολύ πιο ομαλά. Όπως είπε και ο κύριος ε, Καστάλτο, εμείς δεν διαπιστώσαμε σημαίνουσες παρατυπίες ούτε στη διάρκεια της προεκλογικής εξεταρίας ούτε και στη διάρκεια της ε, εκλογικής μάχης την ημέρα των εκλογών. Βεβαίως ε, ε, αυτά πρέπει να τα δει κανείς και υποδοφός και συγκρίνοντας την συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία με την προηγούμενη ακριβώς και τις βελτιώσεις που διαπιστώσαμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φαίνεται ότι οι εκλογές αυτές δεν φαίνεται να ε, ενισχύουν τη διακομματική εμπιστοσύνη στο Μαυροβόνιο γιατί υπάρχει δραματική πόλωση μεταξύ των κομμάτων στο Μαυροβούνιο γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών που θα γίνουν στην Ποτγκόρτζα τον επόμενο μήνα. Παρ' όλα αυτά σημειώνουμε ότι πάνω από το 66% των εκλογέων υποστήριξαν φιλοευρωπαϊκές, φιλοδυτικές δυνάμεις, κάτι που επιβεβαιώνει ότι το Μαυροβούνιο κινείται σε σωστή ε, κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά βεβαίως πρέπει να ε, συνεχίσουμε να ελέγχουμε την κατάσταση, να την, να την ε, παρακολουθούμε, ε, διότι όπως έχουμε πει το Μαυροβούνιο είναι η ναυαρχίδα μεταξύ των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Κύριε Τάνοκ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Φάμπιο Καστάλντο, για την εξαιρετική του παρουσίαση. Εγώ ε, διάβασα και την προκαταρκτική έκθεση που έχει συνταχθεί που συνάδει με αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Καστάλτο. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει το ε, ε, Μαυροβούνιο ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Ο κύριος Τζουκάνοβιτ ε, εντάξει, ευθύνεται για κάποιες, ε, κάποια μικρά παράπονα που ακούστηκαν, αλλά ε, τίποτα το σημαντικό όπως αναφέρεται άλλωστε και στην έκθεση και στις, στην παρουσίαση του κυρίου Καστάλτο. Θεωρούμε ότι ε, επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα του αποτελέσματος ε, του, αυτού του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών. Βεβαίως χαίρομαι πολύ διότι το ζήτημα αυτό μας, με έχει απασχολήσει και μένα ως μόνιμο εισηγητή τα τελευταία 7 χρόνια ε, ήταν, υπήρχε ανάγκη βελτίωσης της νομικής βάσης για την πραγματοποίηση των εκλογικών διαδικασιών στο Μαυροβούνιο. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έχει γίνει. Υπήρχε ευρεία επιλογή υποψηφίων και όπως είπε και ο συνάδελφος Πίτσουλα φαίνεται ότι εκφράστηκε μεγάλη υποστήριξη από τις εκλογές προς ε, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Θεωρώ λοιπόν ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί ένα success story και χαίρομαι για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τζουκάνοβιτς είναι πλέον ένας από τους αρχαιότερους ε, ε ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων που θα έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θυμάμαι ότι ο κύριος Τζουκάνοβιτς για, κάποια, ε, για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα ήταν πρόεδρος του Μαυροβουνίου ακόμα και όταν ήταν ε, ομόσπονδο κρατήδιο της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας στη συνέχεια ήταν πρωθυπουργό για πολλά χρόνια εν πάση περιπτώσει έχει πολύ μεγάλη εμπειρία ο άνθρωπος αυτός γι' αυτό και νομίζω ότι η πρόσκληση από τον κύριο Ταγιάννη προς τον Τζουκάνοβιτς ε, θα ήταν ένα πολύ θετικό δείγμα εμείς πάντως ως πολιτικό ομάδα θα υποστηρίξουμε τέτοια πρόσκληση Ωραία. Όταν μιλούσατε για τις προηγούμενες θέσεις του κ. και ο Σπιτσούλα ε, ε, συγκατένευσε. Έχετε καλή γνώση της ιστορίας της Ιουγκοσλαβίας προφανώς. Άλλα σχόλια. Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Καστάλτο. Προσπαθούμε να πιάσουμε το χρονοδιάγραμμά μας και το στόχο μας. Περνάμε στο σημείο 6. Ε, έχουν έρθει οι καλεσμένοι μας. Good to see you, Ambassador. How are you doing? Περνάμε στο σημείο 6. Συζητούμε το θέμα των τελευταίων επεισοδίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας της ε, Κύπρου και πιο συγκεκριμένα το μπλοκάρισμα ε, των πλοίων που ήταν να κάνουν γεωτρήσεις ε, και τα οποία είχε δώσει άδεια η η Δημοκρατία. Καταρχήν, να καλωσορίσω τον πρέσβη κύριο Νικόλαο Εμιλίου και να καλωσορίσω και την γνωστή μας Αγγελίνα Άικχορστ, ε, αναπληρώτρια διευθύνουσα ε, ε, διευθύντρια της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με αρμοδιότητα Δυτικά Βαλκάνια, Δυτική Ευρώπη και Τουρκία. Η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για, για την εξέλιξη στην Τουρκία με πολλές επικρίσεις για τις εξελίξεις. Επιπλέον, ε, Εκτό τη της ε, εσωτερική κατάσταση, η Τουρκία γίνεται όλο και πιο επιθετική είναι των γειτόνων τη, συμπεριλαμβανομένων και των γειτόνων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια συζητήσαμε το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία. Σήμερα θα συζητήσουμε την, ε, τις ε, τελευταίες ε, δράσεις της Τουρκίας μέσα στην ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Οι τουρκικά πολεμικά πλοία μπλοκάρισαν γεώτρηση που ήταν να γίνει από πλοία της Ιταλικής Ένη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ε, ήταν, αυτό ήταν μόνο το τελευταίο από μια σειρά παρόμοιων ε, επεισοδίων. Ε, η Τουρκία επανειλημμένω έχει μπλοκάρει τέτοιου είδου προσπάθειε γεωτρήσεων στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατα, κατήγγυλαν και καταδίκασαν ρητά αυτές τις δραστηριότητες της Τουρκίας. Ήδη τον Νοέμβριο του 2014 το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα που ενθάρρυνε την Τουρκία να δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει αυτές τις προκλητικές δράσεις στην ε, ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη ε, της ε, Κύπρου. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο, αν θέλεις και εσύ Αγγελίνα, πρώτα στον πρέσβη κύριο Εμιλίου και μετά θα ακούσουμε και την δική σου άποψη. Σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή και για τις ηγετικέ σας παρατηρήσεις, αλλά και για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτηση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και με την κυρία Άιχος, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα σας εκπλήξει αν πω ότι θα ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένος αν σήμερα μπορούσα να σας μιλήσω για την ε, συνεργασία και τις συμπράξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι ε, για τα ε, πρόσφατα γεγονότα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σε τελική ανάλυση, η, Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι προσανατολισμένη στην συνεργασία με όλους τους ε, γείτονές μας. Πιστεύουμε στεναρά ότι η συνεργασία και οι συμπράξεις στον τομέα των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να οικοδομήσει σχέσεις μεταξύ των χωρών της, της περιφέρειας και να ενισχύσουν την σταθερότητα και την ειρήνη. Για το σκοπό αυτό η χώρα μου έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και διμερός αλλά και πολυμερός με τις ε, γειτονικές της χώρες όπως είναι ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ορδανία και η Ελλάδα. Οι σκοποί μας ε, συνάδουν πλήρως με την ενωσιακή στρατηγική που ε, έχει ε, αναδείξει την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγική προτεραιότητα. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των, της ενωσιακής στρατηγικής, της πολυμορφίας και της διαφοροποίησης τόσο των ενεργειακών δρόμων και των ενεργειακών πόρων. Η ανακάλυψη υδρογόνων ανθράκων, κοιτασμάτων υδρογόνων ανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και οι μελλοντικέ ενδεχόμενες τέτοιες ε, ανακαλύψεις μπορούν να συμβάλλουν στην ευημερία και την ασφάλεια της περιοχής. στο πλαίσιο της σύμβασης του ΟΗΕ για τη θάλασσα, η Κύπρος το 2004 ανακήρυξε την ε, δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επιπλέον, εκ έκτοτε έχει υπογράψει ε, συμφωνίες με το Λίβανο, ε, το Ισραήλ και την ε, Αίγυπτο. Δεν έχουμε κρυφή ατζέντα. Σκοπός μας είναι η συνεργασία, η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας οικονομικής και κοινωνικής με όλους τους γειτονές μας μια μορφή συνεργασίας που θα είναι επωφελής για όλες τις χώρες της περιοχές που θέλουν να συμμετέχουν στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της στήριξης του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας των συμμετεχουσών χωρών. Η Κύπρος ε, έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους γείτονές της. Εκτός βεβαίως από μία ε, αξιοσημείωτη ε, εξαίρεση. Κάτι όμως που δεν οφείλεται στη, στην στάση της Κύπρου. Οι τουρκικές ενέργειες στην, στην Κυπριακή ΑΟΣ μας έχουν σκόπο να... Ε, ενισχύσουν και να προωθήσουν τα δικά της συμφέροντα, δηλαδή τον έλεγχο των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ε, μετατροπή της σε κόμβο ενεργειακό ε, στην Ανατολική ε, Μεσόγειο. Ταυτόχρονα εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται οι ενέργειες αυτές αποτελούν ξεκάθαρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πολιτικά και οικονομικά επενδύσει στην προοπτική, την ενεργειακή προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε τεχνικές και ε, οικονομικές μελέτες ε, όσον αφορά τα, τις δυνατότητες της Ανατολικής ε, Μεσογείου για τη μεταφορή, μεταφορά ε, ενέργειας μέσω Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας. Οι δράσεις της Κύπρου ε, συνάδουν πλήρως με ε, οι δράσεις της ε, Τουρκίας ε, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις υποχρεώσεις μιας υποψήφιας χώρους όπως είναι οι καλές σχέσεις γειτονίας και η ειρηνική επίλυση διαφορών. Επίσης παραφιάζουν τις διατάξεις τον, τη, τον, τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005 αλλά και το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Ένα έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι κανόνες του παιχνιδιού και που εθελοντικά η Τουρκία έχει συνυπογράψει και που προβλέπει την εξομάλυνση των σχέσεων της Τουρκίας με όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένες της Κύπρου. Αντιθέτως λοιπόν η Τουρκία επιθετικά ε, έχει σταθεί απέναντι στην Κύπρο και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 23 Μαρτίου το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα ε, δικαιώματά της στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Περνάω τώρα στα πρόσφατα γεγονότα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2018 τουρκικές ναυαρχίδες με την απειλή ε, χρήσης βίας προσπάθησαν να μπλοκάρουν ε, ε, γεωτρύπανα της Ιταλικής εταιρείας ENI, ε, τα οποία είχαν λάβει άδεια για δραστηριοποίηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η πλατφόρμα ε, επρόκειτο να ε, στηθεί 15 ναυτικά μίλια στο οικόπεδο 3 της Κυπριακής ΑΟΣ το, το σχέδιο της ENI ε, είχε λάβει άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία και η πλατφόρμα εξόρυξης απετράπει η κατασκευή της ε, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι η Τουρκία επρόκειτο να εκτελέσει στρατιωτική επιχείρηση με πραγματικά πείρα παρά τις προειδοποιήσεις και τις καταγγελίες της Κύπρου. Πρόκειται για περιοχή την οποία κατέκτησε ε, σκόπιμα η Τουρκία προκειμένου να παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της ε, Κύπρου. Στις 23 Φεβρουαρίου 2018, έπειτα από 13 μέρες τέλματος, οι πλατφόρμες της ENI προσπάθησαν να φτάσουν στο στόχο τους, αλλά και πάλι μπλοκαρίστηκαν από τουρκικά πολεμικά πλοία υπό την απειλή χρήσης βίας. Το περιστατικό αυτό αποτελεί σαφή κλιμάκωση της κυπριακής επιθετικής στρατιωτικής δράσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με στόχο ε, την πραγματοποίηση ακόμη και στρατιωτικών ε, ασκήσεων εντός των ε, χωρικών υδάτων της Κύπρου και στο FIR της. Και φαίνεται σαφώς ότι μέσα από αυτή την παράνομη κλιμάκωση η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα εκφοβισμού για τις εταιρείε που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο στην Κυπριακή ΑΟΣ σε μια προσπάθεια να ε, αποτρέψει την συνεργασία τους με την κυβέρνηση της Κύπρου. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ε, αποκλειστική οικονομική της ζώνη όπως φαίνεται από μια σειρά από ψηφίσματα και δηλώσεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι μεγάλες πετρελομηχανίες έχουν λάβει άδεια για εξόριξη και έρευνες. Η Κύπρος δεν έχει εξαντλήσει ακόμη τα νομικά της δικαιώματα. Είναι γεγονός όμως ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή η επιθετικότητα της Τουρκίας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί βεβαίως με ε, ειρηνικά μέσα και με μέσα δικαιοσύνη. Η Κυπριακή κυβέρνηση επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση προσπαθώντας να επιβάλλει και να ασκήσει τα, κυριαρχη, τα κυριαρχιακά της δικαιώματα ενεργώντας ως σοβαρός εταίρος στην Ανατολική ε, Μεσόγειο και αποφεύγοντας την κλιμάκωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και όλα τα άλλα μεγάλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφήνεια έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ε, Κύπρου. Να υπενθυμίσω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου με τίτλο «Ενέργειες της Τουρκίας που δημιουργούν ένταση στην ε, Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη» του Νοεμβρίου 2014 καθώς και διαδοχικές εκθέσεις του Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και την τελευταία ετήσια έκθεση της Κομισιόν σχετικά με την πρόοδο των ε, ε, διαπραγματεύσεων προσω, προσχώρησης της Τουρκίας. Όλοι οι φορείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν επιβεβαιώνουν ότι οι τουρκικές ενέργειες αποτελούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένων ε, και εκκλήσεων προς την Τουρκία να μην ε, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής ε, Δημοκρατίας και κάνοντας έκκληση προς αυτοσυγκράτηση ε, και καλώντας την να μην απειλεί με τη χρήση βία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στα τελευταία του συμπεράσματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Μαρτίου υποστήριξε και υπογράμμισε την αλληλεγγύη του με την Κύπρο και καταδίκασε τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, κάλεσε την την ε, Τουρκία να σταματήσει τις ενέργειες αυτές, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της ε, Κύπρου, να, να... να πραγματοποιεί έρευνες ε, στα χωρικά της ύδατας σε σχέση με φυσικούς πόρους σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επίσης υπογράμμισε τη σημασία εξομάλυνσης των σχέσεων της Τουρκίας με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μήνυμα βεβαίως δόθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση στη Βάνα στον κύριο Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία επμένει στις θέσεις της ε, και θεωρεί ότι τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα ε, σε αποκλειστική οικονομική ζώνη παρά μόνο σε ε, χωρικά ύδατα. Και βάσει αυτής της παράδοξης άποψης η Τουρκία επιμένει στη δική της θέση και θεωρεί ότι η δική της ερμηνεία του διεθνούς δικαίου είναι σωστή. Επιπλέον η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και τις συμφωνίες περιορισμού αυτών με τους γειτονές της. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ε, υιοθετήσει μια πολύ σαφή ε, θέση λέγοντας ότι και οι Τουρκοκύπροι θα ωφεληθούν από τα κοιτάσματα υδρογονάνθρακων στην προοπτική επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Επίσης, έχει συμφωνηθεί ότι οι υδρογονάνθρακες και οι ενεργειακοί πόροι θα εμπίπτουν στην ε, αρμοδιότητα της ομόσπονδης κυβέρνησης ενώ η εξόριξη, η διερεύνηση κοιτασμάτων ε, επίσης θα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης. Τα έσοδα δε ε, από τους, τους υδρογονάνθρακες θα είναι δυσανάλογα μάλιστα υψηλά για την τουρκοκυπριακή κοινότητα ε, ε, έως ότου καλυφθεί ε, η απόσταση που χωρίζει τις δύο κοινότητες. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας κάτι θετικό. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινώς αποδεικτή βιώσιμη λύση του κυπριακού ζητήματος το συντομότερο δυνατό. Μια τέτοια εξέλιξη θα μετέτρεπε την, τα κοιτάσματα υδρογονανδράκων της Ανατολικής Μεσογείου σε καταλήτη της ειρηνικής συνεργασίας και της ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον Εμίλιο ε, νομίζω κατέληξε σε μια θετική νότα, δηλαδή θα πρέπει να βλέπουμε, το πράγμα, να βλέπουμε τα πράγματα θετικά και να αναζητάμε ευκαιρίες συνεργασίας στην Μεσόγειο. Όπως είπε όμως σήμερα και ο Πρόεδρος και ο κύριος Πρέσβη, το γεγονό ότι είχαμε σχέσεις αντιδράσεις και από το Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο, από την κυρία τα κτλ η οποία ήταν σαφέστατη στι τοποθετήσει της, δηλαδή πλήρης ελεγγύη με την Κύπρο και έκκληση προς την Τουρκία για πάυση παράνομων δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο και το σεβασμό του κυριαρχού δικαιώματος της Κύπρου να ερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς τους φυσικούς, τους, φυσικούς της συγγνώμη, πόρους σύμφωνα με το διεθνές και κοινωνικό δίκαιο. Και όπως είπε και ο κύριος Πεσβευτής, και αυτά τα συζητήσαμε με τον κύριο Ερντογάν στην Βάρνα, το συζητήσαμε σε επίπεδο υπηρεσιών, σε επίπεδο διοικήσεων επανειλημμένως, μεταξύ των διαφόρων επαφών μας με τους εταίρους μα από την Τουρκία και είναι σημαντικό αυτό γιατί ω χώρα υποψήφια Φαίνεται ξεκάθαρα από τις εκθέσεις της Κομισιόν, ακόμα και από την πρόσφατη που ανέφερε ο Πρόεδρος, ως χώρα υποψήφια είναι δεσμευμένη η Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να έχει καλές σχέσεις γειτονία με όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένες και τη Κύπρου. Η κυρία Μογκερίνη λοιπόν και όλοι οι θεσμοί και οι ηγέτες της Ένωσης επανειλημμένως τονίζουν αυτό το στοιχείο ξεκάθαρα ότι είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο, το θέμα των καλών σχέσεων γειτονία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υποψήφιε χώρες όπως την Τουρκία. Και δεν μπορώ παρά να επαναλάβω και εγώ αυτή την έκκληση, δηλαδή για αποφυγή περαιτέρω δράσεων στα πλαίσια της Κυπριακής ΑΟΣ που θα μπορούσαν να βλάψουν τις καλές σχέσεις γειτονίας και θα μπορούσαν να βλάψει και τις σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία και να βλάψει επίσης και την περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή. Είναι λοιπόν τώρα σημαντικό να υπάρξει αποκλιμάκωση, να αναζητηθεί και να βρεθεί μια λύση και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτό και ο κ. Πρέσβης μας ενθαρρύνει το γεγονό ότι οι Κύπροι ηγέτες ατύπως δείπνησαν την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί γιατί τα πλεονεκτήματα από μια τελική λύση υπό την αιγίδα του ΙΕ είναι πάρα πολλά και πρέπει να γίνει μια ολοκλήρωση αυτή της καλής δουλειά που έχει ξεκινήσει. Εμείς ελπίζουμε να και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε επικοδομητικά προς το κοινό συμφέρον όλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ Αγγελίνα Αϊκχόρστ. Ακούσαμε τους προσκαλεσμένους μας, θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Έχουμε υψηλή συμμετοχή από συναδέλφους από την Κύπρο. Μου έχουν ζητήσει να μιλήσουν ο κ. Παπαδάκης, ο κ. Ναυρίδης, ο κ. Θεοχάρους, ο κ. Τάνοκ, ο κ. Χατζηγεωργίου, ο κ. Ηλικιώτης και ο κ. Καστάλτο. Ε, αυτοί όλοι ή μου ξέφυγε κάποιος. οκτώ συνάδελφοι. Δύο λεπτά παρακαλώ στον καθένα. Δίνω το λόγο στον κύριο Παδάκη καταρχήν. Τρία σημαντικά σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι με τη συνεχιζόμενη συμπεριφορά της Τουρκίας οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει στάση να θέλει να πετύχει κάτι. Και εξηγούμε. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαμε να δώσουμε το δόλο μας στην Τουρκία να ανοίξουν τα κεφάλαια για να γίνει πιο δημοκρατική η χώρα. Ανταυτού είδαμε την Τουρκία να γίνεται περισσότερο αυταρχική καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ίδια την Τουρκία εισβολή στο Αφρίν, εισβολή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να συζητήσει σοβαρά για λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας, οικονομικών μέτρων, sanctions, κατά αντίστοιχων τρόπων όπως έγινε με τη Ρωσία. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να ξεπηδήσουν πραγματικά δημοκρατικές δυνάμεις εντός της Τουρκίας. Το συνοχιζόμενο χαίδεμα του κυρίου Ερτογάν αλλά και της αντιπολίτευσης οι οποίοι καθημερινά παράγουν εθνικισμό δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, αντίθετα θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Το δεύτερο σημείο. Οι παραβιάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου είναι παραβιάσεις της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κοιτάσματα στην ΑΟΣ της Κύπρου είναι ευρωπαϊκά κοιτάσματα και μπορεί να είναι εναλλακτική πηγή ενέργειας για την ίδια την Ευρώπη τη στιγμή που εξαρτάται από κάποιους τρίτους. Και το τελευταίο σημείο, να σταματήσουμε τα ευχολόγια, να θεωρούμε ότι το Κυπριακό θα λυθεί μόνο με τις ευχές και Υπάρχουν στιγμές που θεωρώ ότι στην Επιτροπή έχετε λαθασμένη εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά στο Κυπριακό. Όταν η Τουρκία συνεχίζει να θέλει να έχει εγγυητικά δικαιώματα στην Κύπρο, στρατεύματα κατοχής, πώς μπορούμε να κάνουμε αποδεκτή την οποιαδήποτε λύση η οποία θα περιέχει αυτά τα στοιχεία μέσα στη λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Θαγουάρουσα, στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως μας είπε τις προάλλες η κυρία Μογκερίνη δια του εκπροσώπου της αυτού που την αντικαθιστούσε στην Ολομέλεια, η Τουρκία είναι ένας ισχυρός παίκτης στην περιοχή, ένας παίκτης κλειδί ένα ισχυρό οικονομικό σίδερο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η απειλή τη Τουρκία εναντίον τη Κύπρου είναι πραγματική και δεν περιορίζεται από το γεγονό ότι έχει ισχυρέ οικονομικέ σχέσει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και δεν πρόκειται να τερματιστεί με την επίλυση του Κυπριακού, γιατί η επίλυση του Κυπριακού για την Τουρκία σημαίνει τον πλήρη έλεγχο τόσο τη χερσαία όσο και τη θαλάσσια έκταση του νησιού και κατά συνέπεια και ε, φυσικών πόρων της ε, Κυπριακής ε, Δημοκρατίας. Αυτό το έχει κάνει ξεκάθαρο η Τουρκία. Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί από την Θράκη όπου υποδαβλίζει την μουσουλμανική μειονότητα σε όλο το μήκος του Αιγαίου μέχρι το Καστελόριζο. Είναι, έχει θέσει την Κύπρο υπό τον κλειό του πολεμικού στόλου της. Έχει κάνει ό,τι έχει κάνει εναντίον του γεωτρύπανου της «Έννη» και ήδη λίγες εβδομάδες πριν από την σύνοδο του Κρανς Μοντάνα στην οποία όλοι είχαν επενδύσει τόσα πολλά έχει ενισχύσει τον στρατό κατοχής με ε, πολλά ε, πολύ, ισχυρής, ε, ε, πολύ ισχυρά πυροβόλα καθώς και άρματα μάχης τα οποία έχουν δεθεί σε επιθετική διάταξη έξω από τη Λευκοσία. Αν αυτό είναι πολιτική επίλυση του Κυπριακού τότε δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι η πολιτική μη επίλυση του Κυπριακού. Ε, άλλωστε η Τουρκία διο, διολυσταίνει προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις εκλογές της 24ης Ιουνίου θα πεθάνει ο Κεμαλισμός και θα αναβιώσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και άλλο ένα τέρας σαν αυτά που έχουν, έχουμε εκθρέψει μέχρι τώρα από τον Καντάφη μέχρι τον Μουμπάρακ μέχρι τον Σαντάμ θα δείτε να δημιουργείται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χατζηγεωργίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι γενικότερες τοποθετήσεις για το Κυπριακό θα έχουμε στην ευκαιρία στη συνέχεια όταν θα γίνει η συζήτηση της έκθεσης της Κομισιόν για την ε, προοπτική της Τουρκίας και άλλων χωρών. Εδώ μιλάμε για κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έχει παραβιαστεί κατ' επανάληψη από την Τουρκία με ιδιαίτερο γεγονός την παρεμπόδιση γεωτρύπανου της ΕΝΗ όταν πήγαινε για συγκεκριμένη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μιλάμε λαγιάδιστα για παραβίαση στη νότια πλευρά της Κύπρου που αυτό σημαίνει ότι γεωγραφικά η Τουρκία ποτέ δεν θα είχε τη δυνατότητα α, οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης. Υπάρχουν συγκλήσεις γύρω από αυτό το ζήτημα που με την επίλυση του Κυπριακού θα συμβάλλουν προς όφελος και των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Και οι συγκλήσεις αυτές λένε ότι οι θαλάσσιες ζώνες αποτελούν ομοσπονδιακή αρμοδιότητα και προσθέτουν επίσης ότι η κατανομή των εσόδων θα γίνεται από την Ομοσπονδία προς όφελος και των δύο κοινοτήτων. Οι φυσικοί πόροι, συνακόλουθα, γενικότερα οι φυσικοί πόροι αποτελούν ομοσπονδιακή υπόθεση. Ανησυχούμε από το γεγονό ότι υπάρχουν τελευταίω κουβέντε από την τουρκοκυπριακή πλευρά που δείχνουν ε, να μειώνεται σε κάποιο βαθμό το ενδιαφέρον για επίλυση του ζητήματος ε, των εσόδων πριν από τη λύση. Αυτό ε, δεν θα βοηθήσει καθόλου προς την κατεύθυνση του ετούμενου στόχου. Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι η καταδίκη η πραγματική καταδίκη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημερινή συζήτηση το καταδεικνύει των παραβιάσεων της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μου επιτρέπει να ξεχνώ ή να υποβαθμίζω την χλιαρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις συνομιλίες στο Κράμον Μοντάνα. Επ' αυτού θα επανέλθω στη συζήτηση για την έκθεση της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καστάλντο έχει το λόγο δύο λεπτά. Πρώτα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε πολύ συχνά στη, για την Τουρκία στην Ομέρια και στην Επιτροπή, αλλά ποτέ θετικά ή έστω ουδέτερα. Και αυτό από μόνο του θα έπρεπε να αρκέσει για να καταδείξει την κατάσταση του τωρινό μα σχέσεων με την Τουρκία. Η σημερινή συζήτηση αφορά ιδιαίτερα την διαχείριση τη Κυπριακή ΑΟΣ, δηλαδή αυτή την θαλάσσια περιοχή όπου το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Ή τουλάχιστον οι γείτονές του θα πρέπει να το αφισβητούν αυτό. Η Τουρκία δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να κρύψει τις επιδιώξεις της για τα κοιτάσματα. Και μέχρι τώρα έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αποτροπή της προσέγγισης μεταξύ δύο κοινοτήτων του νησιού. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει τη στάση αυτή, θα πρέπει να σταματήσει να δημιουργεί εντάσεις και θα πρέπει να μην συμβάλλει αρνητικά σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε ποια είναι τα α, γεγονότα. Ξέρετε για αυτό το γεωτρύπανο τη Έννη, το οποίο απειλήσαν τουλάχιστον τρία τουρκικά πολεμικά. Αυτό το γεγονός είναι μόνο το τελευταίο σε, μια, σε ένα μακροσκυλή κατάλογο πολεμοχαρών δράσεων της Τουρκίας στην Μεσόγειο. Πρέπει να επιθυμήσουμε λοιπόν ότι η η αφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και ο εκφοβισμό, απλά και μόνο αποτελεί ένα κάζους μπέλι για την νομιμότητα. Και μέχρι τώρα έχει προκαλέσει μόνο ρηματικές διακοινώσει από την ε, Ένωση όσον αφορά τη δραστηριότητά της. Η, η ατζέντα, το θεματολόγιο του κυρίου Ερντογάν δεν ε, σταματάει σε αυτό. Έχει περάσει και στην σύλληψη των δύο στρατιωτών και σε άλλα θέματα. Θα έχουμε στη συνέχεια την έκθεση του κυρίου Χάν για τη διεύρυνση. Φοβάμαι ότι όπως συνήθως θα ακούσουμε ότι δεν θα ανοίξουν τα κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις επειδή δεν υπάρχουν πρόοδοι. Η αλήθεια είναι πια ότι η Τουρκία έχει εγκαταλείψει πλήρως την ευρωπαϊκή της πορεία. Και λόγω ακριβώ τη μετανάστευση, εμεί συνεχίζουμε να καθυστερούμε, να χρονοτριβούμε χωρί να υπάρχουν σαφή δείγματα. Αυτή η Τουρκία η Τουρκία δεν θα πρέπει πια να θεωρείται χώρα υποψήφια. Ας αναζητήσουμε κάποια κανάλια συνεργασίας αλλά κυρίω πρέπει να λάβουμε σοβαρά και αποτελεσματικά μέτρα στις ημερεί σχέσεις γιατί η αδυναμία ποτέ δεν οδήγησε σε κάτι το θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Επιτίδιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με όλα όσα έχουν αναφερθεί από τους προλαλήσαντες και την ε, προλαλήσασα ε, συνάδελφο αλλά και αυτά τα οποία γνωρίζει και η Επιτροπή αλλά και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όχι όμως μόνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, παράλληλα προκαλεί και την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία διαφορεί. Συνεπώς, με την όλη συμπεριφορά της η Τουρκία ουσιαστικά έχει θέση εαυτήν εκτός της ευρωπαϊκής προοπτικής. Αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πρώτη που θα το αναγνωρίσει και θα συμπεριφερθεί ανάλογα. Δεν έχει νόημα να διαπραγματεύεται με την Τουρκία όταν η Τουρκία κρατά υπομοιρία την Κυπριακή Δημοκρατία έχοντας στρατεύματα κατοχής δεν της επιτρέπει να ασκήσει κυριαρχικά τις δικαιώματα και επιπλέον εμπέζει και προκαλεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμπεριφορά που επέδειξε πρόσφατα σε ό,τι αφορά το γεωτρύπανο της Έννη. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε πραγματικά να επιλύσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε συνομιλία με την Τουρκία. Να γίνει σαφές στην Τουρκία ότι δεν έχει καμία σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία θέση και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να βρούμε κάποια άλλη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να κινηθούν οι διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Διαφορετικά, όταν εκδηλώνουμε αδυναμία ή φοβία απέναντι στην Τουρκία, θα είμαστε συνεχώς στο σημείο να συζητάμε και να επαναλαμβάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα διάλογο κοφών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτήδια. Ο κύριος Μαυρίτης. Ευχαριστώ πολύ. Αυστηρά στο θέμα, προσδοκώντας να πάρω συγκεκριμένες απαντήσεις ή τοποθετήσεις. Καταρχήν να πω ότι δεν συμμερίζομαι, μακάρι να μπορούσα να συμμεριστώ, την αισιοδοξία που εκφράστηκε έστω κατά κάποιο τρόπο από τον πρέσβη της Κύπρου και εν μέρη από το External Action. Όμως, συμμερίζομαι πλήρως όσα επί της ουσίας τοποθετήθηκαν από τον μόνιμο αντιπρόσωπο. Το ερώτημα όμως για όλους μας και προς τους δύο είναι το εξής. Έχουμε πλήρη στήριξη από όλα τα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα προς τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον κυριαρχικό της δικαίωμα, το οποίο επιβεβαιώνουν τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία. Δεν νομίζω μπορεί να πάει πιο καθαρά υποστηρικτική θέση από αυτό που έχουμε. Άρα το ερώτημα είναι πολύ απλό. Τι είναι το επόμενο που θέλουμε. Θέλουμε ακόμα ένα ψήφισμα, ακόμα μια δήλωση. Αυτό είναι και για τους δύο σας. Και για την Κυπριακή Κυβέρνηση και για την Επιτροπή. Το δεύτερο μου ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον όλοι μας έχουμε αποφασίσει ότι ο τρόπος που ενεργεί η Τουρκία είναι παράνομος και πλήττει τα συμφέροντα και τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, η Ευρωπαϊκή, έγινε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνο για soft issues. Τι είναι τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν για να επιβάλλουμε κυρώσεις. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλουμε ξανά και ξανά κυρώσεις και εδώ δεν βγαίνει καν από το στόμα μας. Αυτό και για τους δύο σας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω κύριε Πρέσβη. Όπως γνωρίζετε, ως ε, φίλος της Κύπρου και της μεγάλης ε, κυπριακής παρικίας που έχουμε στην ε, Βρετανία, χάρηκα πάρα πολύ πριν κάποια χρόνια όταν έγινε η ανακάλυψη των κοιτασμάτων και ιδίως με την ε, προοπτική συνεργασίας και με εταίρους όπως είναι το Ισραήλ. Η Κύπρος πραγματικά αποτελεί ένα success story έπειτα από την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, και θεωρώ ότι η ανακάλυψη αυτών των κοιτασμάτων θα μπορούσε να της δώσουν μεγάλο πλεονέκτημα και για την ευημερία της και για την ενεργειακή ασφάλεια και ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε Άλλωστε υποσχεθεί ότι ο πλούτος αυτός θα μοιραστεί γενναιόδωρα με τους Τουρκοκύπριους εφόσον γίνει η επανένωση του νησιού ε, υπό μία σημαία και ελπίζω οι συνομιλίες να ξαναξεκινήσουν σύντομα. Αυτό είναι, λοιπόν, είναι ένα από τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραβίαση της Τουρκίας και της ε, Κυπριακής αός από την πλευρά της Τουρκίας δηλαδή και την, τις ενέργειες που ε, ανέλαβε ενάντια στο γεωτρύπανο της Ένη ε, και την παραβίαση δηλαδή του δικαιώματος της Κύπρου να συνάπτει εμπορικές ε, σχέσεις. Οι τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας και απέναντι στους γκιουλενιστές, τις μαζικές συλλήψεις αλλά και την αγορά S400 από τη Ρουσία πραγματικά μας ανησυχούν πολύ ε, γενικώ επιδίδεται σε ε, αμφιλεγόμενες ε, ενέργειες και στη θάλασσα η Τουρκία και θεωρώ και εγώ, όπως είπαν και άλλοι, ότι πραγματικά δεν αξίζει η Τουρκία πλέον να θεωρείται υποψήφια προς ένταξη χώρα. Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω λοιπόν εκ μέρου του ECR να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με την Κυπριακή Δημοκρατία και να ευχαριστήσω όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στεναρή στάση που έχουν επιδείξει καταδικάζοντα και καταγγέλλοντα την επιθετικότητα τη Τουρκία και την ε, παρεμπόδιση της ε, Κύπρου να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην ΑΟΣ τη. Ευχαριστώ. Τέλο ο κύριο Σιλικιώτη. Ε, πρώτα απ' όλα να επαναλάβω αυτό που είπε, που είπε και ο πρέσβη, αλλά και άλλοι συνάδελφοι ότι η Τουρκία ε, με τι παράνομε ενέργειε θα έλεγα τι πειρατικέ ενέργειε, παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο, το δίκαιο τη θάλασσα, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακή Δημοκρατία, παρεμπόδισε μια ευρωπαϊκή εταιρεία, διότι η Ιταλική είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία συνήψε συμβόλαια με την Κυπριακή Δημοκρατία την εκμετάλλευση ε, των κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα οποία πραγματικά τα κοιτάσματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Έχουν γίνει δηλώσει, πάθηκα θέσει από όλα τα θεσμικά όργανα που καταγγέλνουν αυτή την παρόνομη δράση τη Τουρκία. Είναι μια έκφραση υποστήριξη και αλληλεγγύη προ την Κυπριακή Δημοκρατία από μέρου τη Ένωση. Είναι σημαντικά και επιβεβλημένη. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε την παράνομη και προκλητή δράση τη Τουρκία. Είναι γι' αυτό που χρειάζονται να ληφθούν ακόμα πιο αποφασιστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ ποια κατευθύνση. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αναφέρθηκε ο συνάδελφο Ζωτάκη, οι ανησυχίε των Τουρκοπρίων καλύπτονται μέσα από τι συγκλήσει που επιτεύχθηκε μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του φυσικού αερίου ε, μετά την λύση και είναι σημαντικές αυτές οι συγκλήσεις οι οποίε ο Γενικό Γραμματεία του ΙΟΣ στην έκθεσή του το Σεπτέμβρη κάνει αναφορά στη σημασία αυτών των συγκλήσεων και περιλαμβάνει και τις, ε, ε, αυτές για το φυσικό αέριο. Εκείνο που χρειάζεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει σε δύο κατευθύνσει. Πρώτα-πρώτα να συνετίσει την Τουρκία με αφασιστικά μέτρα, αλλά και δεύτερον να συμβάλλει ώστε να επαναρχίσει ένα ουσιαστικό διάλογο. Διότι πραγματικά οι φυσικοί πόροι στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να λειτουργήσουν για την ευρύτερη ως παράγοντας ενίσχυσης της ειρήνης, της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή που είναι από τις πιο ε, εμπόλεμες στην πλανήτη μας, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτης για τη λύση του Κυπριανού και την επανένωση της ε, Κύπρου και του λαού Ευχαριστώ. Ωραία. Συναδέλφοι, πολλά τα ερωτήματα που τέθηκαν. Νομίζω ότι τα περισσότερα απευθύνονταν στην κυρία Αντελίνα Άιχορστ, οπότε θα πρότεινα να δώσω το λόγο σε εκείνη πέντε λεπτά και μετά για άλλα πέντε λεπτά στον πρέσβη Εμιλίου και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα θέματα και τις παρατηρήσεις. Θέλω και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, από πολιτική άποψη ήταν πολύ σημαντικό το γεγονό ότι ακούστηκε το ίδιο μήνυμα από όλα τα θεσμικά όργανα σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο και τις θέσεις της σε αυτό το θέμα και αυτό θα παραμείνει έτσι. Και όπως είπα, αποστήλαμε το μήνυμα αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια στους εταίρους μας στην Τουρκία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όπως γνωρίζετε αν εξετάσουμε τις ευρύτερες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και όπως είπε ο κύριος Τόνακ αυτό είναι ένα θέμα που δεν, ε, δεν είναι μόνο το, το θέμα που συζητούμε σήμερα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που μας απασχολούν σε σχέση με τη σχέση μας με την Τουρκία. Βεβαίως ε, έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση αρκετές φορές στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εδώ βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο, στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών. Σε, όποιο, σε όλα τα επίπεδα η Τουρκία ε, αποτελεί υποψήφια προς ένταξη χώρα. Είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να έχουμε σχέσεις με τη χώρα αυτή ε, όπως έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Και αυτό που προσπαθούμε να βρούμε εδώ είναι πραγματικά λύσεις που, στα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Όσο λοιπόν η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα, δεσμεύεται από το σύνολο των κανόνων που δεσμεύουν τις υποψήφιες χώρες. Και καλούμε την Τουρκία να, να τηρήσει τους κανόνες αυτούς. Και αυτό είναι το μήνυμα όλων των θεσμικών οργάνων. Ακούω κάποιοι να ε, λένε ότι θα θέλαμε να πάνε τα θεσμικά όργανα λίγο παραπέρα. Όπως είπα, ε, εμείς ε, στις συζητήσεις μας και στις συζητήσεις της κυρίας Μογκερίνη σε αυτό επιμένουμε. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την Τουρκία αλλά και να είμαστε σαφείς για το ποιες είναι οι δικές μας θέσεις. Ε, ρωτήθηκα γιατί δεν είχαμε ε, σαφέστερη θέση για τις συνομιλίες της Να Ξέρετε ότι η κυρία Μογκερίνη ήταν εκεί, ε, ήταν και ο κύριος Γιούγκερ παρόν. Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και ο ρόλος ο δικός μας είναι να ενθαρρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο και τις δύο πλευρές εξακολουθώ και ξαναβλέπω μάλλον το δελτίο τύπου ε, που είχε εκδοθεί ε, από τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακιντσί ε, όπου αναφέρεται ρητός ότι εντοπίσαμε τις διαφωνίες μας και συνεχίζουμε τις συνομιλίες μας. Αυτό είναι ένα στοιχείο ενθαρρυντικό, γιατί μόνο μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορούμε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχέσεις μας και στην πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία είπα πράγματι, είπα ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων κύριο Ακιντσί. Έχετε δίκιο. Can you use Συγγνώμη, δεν έχουμε δύο προέδρους στην Κύπρο. Έχουμε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγέτη των ε, ανθρώπων που ζουν στα κατεχόμενα. Δεν ξέρουμε αν είναι Τουρκοκύπροι ή αν είναι έπικοι από την υπηρετική Τουρκία. Αναφέρθηκα στη συνάντηση που έγινα και στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε έπειτα από τη συνάντηση αυτή, όπου και οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι ε, διαπιστώσαμε, εντοπίσαμε τις διαφωνίες μας και υπάρχει προθυμία να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτών. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία υποστηρίζουμε, ενθαρρύνουμε και ελπίζουμε να στεφθεί με θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Άιχος, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν εξέφρασα ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία για τις προοπτικές λύσεις. Απλώς διαπιστωτικά είπα ότι ως υπαρκτό γεγονός σε περίπτωση που υπάρχει λύση, τότε οι φυσικοί πόροι μπορεί να χρησιμεύσουν ως καταλήτης για τη συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω όπως το έπραξα και στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, ότι η κυβέρνηση δεν είναι ευχαριστημένη με τις αναφορές της Επιτροπής στην έκθεση προόδου της Τουρκίας σχετικά με το τι συνέβη στο Κράν Μοντανά. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε σαφώς να πει τα πράγματα με το όνομά της και να υπογραμμίσει τον ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε η Τουρκία και ο οποίος δεν ήταν καθόλου υποβοηθητικός σε θέματα που αφορούσαν κυρίως την Τουρκία, δηλαδή τις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού, τα στρατεύματα και τις εγγυήσεις, έτσι τεινάζοντας την διαδικασία στον αέρα. Επίση, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής από την αλληλεγγύη την οποία επέδειξαν οι εταίροι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά δεν αποκλείει το γεγονός να ζητήσει και επιπλέον μέτρα ως επίδειξη αλληλεγγύης αναλόγως των εξελίξεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Okay. Thank you. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας και την κυρία Άχος και τον κύριο Μιλίου και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Δεν βλέπω άλλα σχόλια. Οπότε πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξή μας. Γεια σας, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλά να τα περνάτε, λέει ο Πρόεδρος. Enjoy your life, είπε. Κοινή εξέταση των σημείων 7 και 8. Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελώτη αφενός και της Δημοκρατίας του Ιράκ. Ήδη το Κοινοβούλιο έδωσε την εγκρισή του για τη σύναψη αυτής της Συμφωνίας εταιρική σχέση λόγω όμως της απόφασης του δικαστηρίου χρειάστηκε να τροποποιηθεί η νομική βάση, οπότε χρειάστηκε να ξαναδώσουμε νέα έγκριση βάσει της νέας νομικής βάσης. Φαίνεται ότι το, ζήμα, το θέμα είναι κάπως, συγγνώμη, το ζήτημα είναι κάπως περίπλοκο, οπότε θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Σαΐφη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε κι εσείς, μετά από μια τροποποίηση τη νομική βάση θα πρέπει για άλλη μια φορά να εγκρίνουμε τη Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ιράκ. Και για να το κάνουμε αυτό έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε κάποιε προτεραιότητε στην ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ιράκ. Η δημοσίευση και η έγκριση μια κοινή στρατηγική για το Ιράκ το Γενάρη, όπως επίσης και η δέσμευση των ευρωπαϊκών οργάνων και των χωρών στην διάσκεψη του Κουβέιτ το περασμό Φλεβάρι, θα πρέπει όλα αυτά να μετατραπούν σε συγκεκριμένε αυτέ πράξει υπέρ αυτή της χώρας. Γι' αυτό η Συμφωνία Τρική Σχέση είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο θα οδηγήσει στην ανοικοδόμηση, στη σταθεροποίηση και στη συμφιλίωση τη χώρα. Στην έκθεση αυτή λοιπόν έχω εντοπίσει τις προτεραιότητες της βραχυπρόθεσμες όσον αφορά την δράση της Ένωσης στο Ιράκ. Στου επόμενου μήνες είναι απαραίτητο η Ένωση και οι χώρες μέλη να διατηρήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια την οποία παρέχουν αυτή τη στιγμή, ώστε να βοηθηθούν όλοι οι Ιρακινοί. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πρόσφατα απελευθερωθήσεις περιοχές και κυρίως στις επενδύσεις για την ανοικοδόμηση και δημιουργία πρωτοβάθμιων μορφών υποδομής για είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, επήγει η συμφιλίωση της Ιρακινής κοινωνίας με τη συνέχιση ενός ε, επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και των αρχών του Ιρακινού Κουρδιστάν και πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να γίνει σεβαστή η διαφορετικότητα της χώρας και των τσινστοσών και στατικών της Ιρακινής κοινωνίας ώστε να διασφαλιστεί η ακυρεότητα τη επικράτειας τη χώρα. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα πολιτικό διάλογο στο Ιράκ ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ε, κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα των γυναικών. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί βεβαίω η διαφθορά και θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνη. Επίση θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την τρομοκρατία. Θα πρέπει να έρθει υπόψη η νομολογία η διεθνή νομολογία και ε, θα πρέπει να καταρριφθεί βεβαίω και η θανατική ποινή. Αυτή η, εταιρική, η συμφωνία εταιρική σχέση βεβαίω ανοίγει ένα νέο πλαίσιο συνεργασία σε διάφορου τομεί όπω η εκπαίδευση, η ενέργεια ή ακόμα και η μετανάστευση. Στην έκθεσή μου χαιρετίζω την αποστολή της Ένωσης για τα θέματα ασφάλειας στο Ιράκ. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια αμερόληπτη αστυνομική δύναμη που θα διασφαλίσει την ασφαλεία των πολιτών. Θα πρέπει όλα αυτά να διασφαλίζονται βεβαίω και να συνοδεύονται από απαραίτητε κοινωνικέ και οικονομικέ πολιτικέ που θα ωφελούν όλου του πολίτε του Ιράκ. Η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει το Ιράκ σε όλε τι διαφορετικότητέ του που αφορούν την οικονομία, ώστε να διασφαλιστεί μια βιώσιμη μορφή ανάπτυξη η οποία θα μπορέσει να προκαλέσει, να δημιουργήσει μάλλον θέσει εργασία κυρίω για του νέου ώστε το κοινοβούλιο μα να συμβάλλει με πραγματική προσταμιαξία αξία στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ιράν, ιδιαίτερα διαμορφώνοντας προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν τι δυνατότητε του Ιρακινού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Ms. Ευχαριστώ κυρία Σαΐφη. Περνάμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Φρόιτ, Ράιμοντ, Κόζο και Καστάλτο. Κάποιος άλλος μήπως επιθυμεί το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Τρία λεπτά το πολύ ο καθένας. Θα εξηγήσουμε τον κύριο Φρόιτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Θα πρέπει να αυτοσχεδιάσω κάπως γιατί πριν από λίγα λεπτά έμαθα ότι θα πρέπει να αντικαταστήσω την κυρία Γκόμες η οποία δυστυχώς απουσιάζει. Αν ήταν όμως εδώ, θα είχε, φαντάζομαι σίγουρα, ευχαριστήσει την συγγήτρια την κυρία Σαΐφη για τη θαυμάσια δουλειά το οποίο κάνω και εγώ βέβαια. Το Ιράκ παραμένει ακόμα σε μια φάση μαθησιακή όσον αφορά τη δημοκρατία. Πριν από 15 χρόνια ε, τέθηκε τέλος στη δικατορία του Σαντάμ μετά από περίοδο εξουσίας ενός τετάρτου του αιώνα με πολλή βία. Αν δούμε βέβαια και το τι έγινε στην Συρία, θα καταλάβουμε ότι το Ιράκ έχει κάνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την θεσμαθέτηση δημοκρατικών θεσμών. Παραδείγματο χάρη, έχουμε τις, ε, είχαμε τι επερχόμενε ε, εκλογέ του Μαΐου και ελπίζουμε ότι από αυτέ τι εκλογές οι τρεις κύριες ομάδες, Σουνίτες, οι κούρι θα καταφέρουν να συνεργαστούν για να ενισχύσουν τη δημοκρατία και να ενισχύσουν το κράτος δικαίου ώστε να αποφελεθούν των επιδευμάτων τους, των προσφάτων. Ένα από αυτά είναι το ότι το, το Ιράκ κατάφερε να συνεργαστεί με τη Σαουδική Αραβία αφενός και με το Ιράν αφετέρου και επιπλέον διατηρεί καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ ή για να το πούμε πιο ειλικρινά οι ΗΠΑ διαδραματίζουν ακόμα ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή και στην πρόοδο των δημοκρατικών θεσμών του Ιράκ. Συνεχίζουμε να καλούμε το Ιράκ βεβαίως να καταπολεμήσει την διαφθορά και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο πλαίσιο αυτού ζητούμε την κατάργηση της θανατικής πηγής. Ποινή, συγγνώμη. Ελπίζουμε λοιπόν μετά τη διεξαγωγή των εκλογών να συνεχίσουν να συνεργάζονται το Ιράκ και η Ένωση ώστε πραγματικά να μετατραπεί σε μια ειρηνική και αναπτυγμένη χώρα του Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Ράιμον για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Χαιρετίζουμε το σχέδιο έκθεση. Θεωρούμε ότι αναφέρεται στα σωστά σημεία και θέματα, ιδίως όσον αφορά την ε, σημασία της διαφορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το IDP. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει και να υποστηρίξει όλες αυτές τις προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος ε, δικαίου, τι ε, θρησκευτικέ διαιρέσει στο Ιράκ ε, χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ κεντρικής ε, κυβέρνησης και τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πρέπει επίσης να κατευθύνουμε προσπάθειες και χρήματα ως Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα εκεί, ιδίως ε, στις παράκτης περιοχές. Και γι' αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων φορέων στην επερχόμενη διαδικασία ανοικοδόμησης. Ε, επίσης, μας χαροποιεί η αναφορά που γίνεται στην έκθεση σε μειονότητες. Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε αυτή την αναφορά και με αναφορά στις ε, θρησκευτικές διαιρέσεις που υπάρχουν στο Ιράκ και την ανάγκη υπέρβασης αυτών. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει ζωτικό συμφέρον να ξεπεραστούν αυτές οι διαιρέσεις ε, και να καταλήξουμε γενικά σε ένα θετικό κείμενο. 1,5 λεπτό λοιπόν χρειάστηκα πρόεδρε, νομίζω δεν χρειάζεται να τα εξαντλήσω και τα δύο λεπτά που μου δώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούζο έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε με την συμφωνία αυτή που περιλαμβάνει σημαντικά τμήματα όπως ε, συμφιλίωση, ενίσχυση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ και κυρίως προσπάθεια αντιμετώπισης των τεραστίων επιπτώσεων της εισβολής που προκάλεσε πάνω από ένα εκατομμύριο νεκρούς. Εμείς ήδη είπαμε παλαιότερα κάτι σε σχέση με τους ε, καθολικούς και την εκδίωση, εκδίωξη των χριστιανικών και όχι μόνο κοινοτήτων αλλά και των εβραϊκών. Έχουμε γύρω στις, στα 78 δόγματα θρησκευτικά στην χώρα, οπότε θα πρέπει να αναφερόμαστε όχι μόνο στους ε, χριστιανούς, αλλά στους Σουνίτες, στους Ιήτες και σε όλα τα θρησκευτικά δόγματα τα οποία διώκονται. Με αυτή την προσέγγιση νομίζω θα βοηθηθεί πολύ το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κ. Καστάλτο για το ε, EFTD. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κ. Σαΐφη για τα μάσκα δουλειά που έκανε. Πολύ πλήρη η έκθεση και συμφωνώ για το γεγονό ότι περισσότερο από ποτέ είναι τώρα απαραίτητο να στηρίξουμε τι δρακινέ αρχέ στην φάση ανοικοδομή τη χώρα. Μια μικρή παρατήρηση. Συνειδητοποιούμε το ότι το ακόμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει πάρα πολλέ προκλήσει σε επίπεδο θεσμικό, διοικητικό, σε επίπεδο κράτου δικαίου και σε βαθμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έλλειψη ενός ισχυρού κράτους τα τελευταία χρόνια ενίσχυσε αρνητικά την διαμάχη των εξουσιών, μάλλον τη μάχη για την εξουσία μεταξύ των διαφόρων φατριών. Οπότε πρέπει όλες οι παρούσες κοινότητες στο Ιράκ να εκπροσωπηθούν εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 12 η Μαΐου υπέρ του συνόλου του πληθυσμού του Ιράκ. Είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μετά ISIS, να ενισχύσουμε όλες τις προσπάθειες οι οποίες αποβλέπουν σε μια πραγματική εθνική συμφιλίωση και μια δίκαιη δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει τα τραύματα που προκάλεσε το Ισλαμικό κράτος. Μέσω λοιπόν των συμφωνιών συνεργασίας θα πρέπει να δείξουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε τη δημιουργία υποδομών, σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Κάτι που θα βεβαίως θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους Ιρακινούς, αποφεύγοντας ε, το κίνδυνο ε, στρατολόγησης από εξτρεμιστικές ομάδες, αλλά κυρίως θα πρέπει να ενισχύσουμε τις διάφορες αρχές της χώρας προς κοινωνικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την σταθεροποίηση της χώρας και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση, η οποία θα, πρέπει να έχει πολιτικές περιεκτικές, δημοκρατικές και η οποία θα διασφαλίσει την πλήρη και δημοκρατική εκπροσώπηση στις μορφές εξουσίας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι ελλείψεις αυτού του είδους θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των τσιχαντιστών και σε στρατολογήσεις. Και αντιθέτως και αντιστρόφως με την πλήρη ενσωμάτωση όλων των συνιστοσών της κοινωνίας θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε αυτό το κίνδυνο. Ευχαριστώ για μια φορά την συγκέντρια θαυμάσια δουλειά της. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Καστάλτο. Ένας ομιλητής έχει συζητήσει το λόγο, ο κύριος Τσάρλς Τάνοκ. Θα είμαι τηλεγραφικός, πρόεδρε. Η ομάδα μου στηρίζει την έκθεση και τις συστάσεις ε, ως πρόεδρος της ομάδας φιλίας με το Κουρδιστάν θα ήθελα να καλωσορίσω τα σχόλια που γίνονται για την επανεκκίνηση του διαρθρωμένου διαλόγου με τις αρχές της Ερμπίλ. Ιδιαίτερα σε, επίσης καλωσορίζω την ε, έκκληση να ξαναρχίσουν οι κατευθείαν πτήσεις ε, προς το Κουρδιστάν που είχαν διακοπεί. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 13, ε, στο Βρετανικό τύπο δημοσιεύτηκε ένα τρομακτικό άρθρο για κάποιες δίκες που έγιναν εναντίον γυναικών μαχητών του Ισλαμικού στρατού, οι οποίες, πολλές από τις οποίες καταδικάστηκαν σε θάνατο, χωρίς να έχουν οι ίδιες διαπράξει κλίματα πολέμου. Πολλές φορές κατηγορούνταν ακόμα και τα παιδιά τους. Πολύ συχνά οι κατηγορίες περιορίζονταν στο ότι ήταν γυναίκες ή παντρεμένες ε, με μαχητές του Ισλαμικού στρατού. Καταλαβαίνω γιατί αυτό στο Ιράκ ε, θεωρείται τρομακτικό, δεδομένου ότι οι ίδιοι μαχητές διέπρεξαν τη δεχτή εγκλήματα. Το γεγονό όμως ότι υπάρχει περίπτωση ε, νέες γυναίκες να... Ε, ε, καταδικαστούν σε θάνατο και να εκτελεστεί η θανατική ποινή μόνο επειδή είναι γυναίκες μαχητών. 12 από αυτές μάλιστα είναι και τουρκάλες, δεν είναι καν Ιρακινές, χωρίς ε, κανενός είδους στοιχείο διάπραξης εγκλήματος. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο ακούγεται καλά σε εμά. Νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους διεθνώς. Είναι σαφές ότι είναι σαφή τα, τα εγκλήματα ε, του Ισλαμικού κράτους ε, και δεν είμαι πολύ σίγουρος ούτε εγώ, ίσως ούτε η κυβέρνησή μου αν θα θέλαμε αυτοί οι μαχητές να έρθουν στη Βρετανία παράδειγμα να δικαστούν ή θα πρέπει να δικαστούν επί τόπου αλλά αυτές οι γυναίκες να κατηγορούνται και να καταδικάζονται μόνο και μόνο επέλεξαν να παντρευτούν κάποιον από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε ε, θέλετε να πείτε δύο λόγια. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα τους τα σχόλια. Σημείωσα τις παρατηρήσεις τους. Πιστεύω ότι συμφωνούμε πως το Ιράκ θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ενισχύσουμε χωρίς καθυστερήσεις τη συνεργασία για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ε, θα συνεχίσω να συζητώ με τους ε, και θα εξετάσω προσεκτικά τις τροπολογίες που έχετε υποβάλει. Ευχαριστώ. Good, thank you. The timetable. The deadline for the amendments is for 20... Τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 26 Απριλίου, 11 το πρωί. Ε, στις 7 Ιουνίου θα συζητηθεί στην ε, ε, Επιτροπή, στις 20 ψηφοφορία και στην Ολομέλεια πριν την καλοκαιρινή διακοπή. ενδεικτικά όλα αυτά. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ανταλλαγή απόψεων με τον Δανιέλε Βιώτη, εισηγητή για τον προπολογισμό της Επιτροπής του 2019. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο κύριος Βιώτη, ε, κύριε Βιώτη είναι εισηγητής για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής του 2019, τον επόμενο χρόνο δηλαδή. Όπως κάθε χρόνο η Επιτροπή μας θα υιοθετήσει γνωμοδότηση και θα ψηφίσει για τις δημοσιονομικές τροπολογίες τον Αύγουστο ε, στο κεφάλαιο, ε, στον τίτλο 4 του πολιτισμού νομικού πλαισίου βρίσκεται η υπηρεσία εξωτερικής δράση. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. ορίζω τον κύριο Βιώτη και μετά τον κύριο Μπενιφέ που είναι ο εισηγητή τη νομοδότης ΑΦΕΤ για το θέμα αυτό. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σα που με φιλοξενεί. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο για να ακούσω και τις απόψεις του εισηγητή σα και των σχεδόν σα. Γιατί σε γενικές γραμμές πρέπει να τονίσω ότι βούλησή μου είναι το να υπάρχει ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα είναι αποδεκτός από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων αλλά και των επιτροπών και ότι θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους που θα με βοηθήσουν στη σύνταξη του προπολογισμού του χρόνου, και ιδιαίτερα στη φάση της συνδιαλλαγής. Σύντομα να αναφερθώ στο θεματολόγιο θέματα στα οποία επικεντρωθήκαμε στις κατευθυντήριες γραμμές που υποβάλαμε και ψηφίσαμε το Μάρτι στην Ολομέλεια. Αναμένω και ενδείξεις από εσά. Καταρχάς, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και να δουλέψουμε σκληρά για το εργαλείο που αφορά τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Όπως ξέρετε, αποφασίστηκε να πάμε στο δεύτερο σκέλος της των κονδυλίων, δηλαδή τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα είναι πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε αυτά. Και σήμερα και σε αυτό συμφωνούμε η Κομισιόν προτίθεται να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, δηλαδή το 1 τρίτο θα προκύψει από τον κοινωνικό προπολογισμό και τα 2 τρίτα θα προκύψουν από τη χρηματοδότηση των χωρών μελών. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί απολύτως με αυτό βέβαια η πιο αρνητική αντίδραση κάποιων χωρών μελών λέει να χρηματοδοτήσουμε πλήρως αυτό το εργαλείο για τους ε, πρόσφυγες στην ε, Τουρκία με χρήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό θα οδηγήσει σε περικοπές άλλων κονδυλίων και δαπανών και επενδύσεων που παραδοσιακά κάνουν το Κοινοβούλιο και η Ένωση. Και αυτό βεβαίω θα ήταν πολύ ανησυχητικό για όλου μας και για τις πολιτικές μας που εδώ και χρόνια εφαρμόζουμε. Δεύτερο θέμα για το οποίο θα πρέπει να δεσμευτούμε είναι οι προκλήσεις για την ασφάλεια και ιδιαίτερα η πρόσφατη πρωτοβουλία της Κομισιόν για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα της άμυνας ως πρώτη φάση δηλαδή ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Άμυνα. Εμείς στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει αποκλειστικά να χρηματοδοτηθεί με ειδικά κονδύλια και όχι μέσω ανακατανομής των υπαρχόντων κολυδίων στα υπάρχοντα προγράμματα, γιατί αυτό προφανώς σημαίνει περικοπές για τα υπάρχοντα προγράμματα. Άλλα τρία-τέσσερα θεματάκια πάνω στα οποία θα πρέπει να δουλέψουμε. Η βελτίωση της στήριξη για την κοινωνία και στην Ανατολή αλλά και στη Μέση Ανατολή και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης που αφορά θέματα ασφάλειας θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την Ούρβα, δηλαδή το εργαλείο στήριξης του Παλαιστινιακού λαού. Υπήρξε μια απόφαση εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης να μην συμβάλλουν πια στον προπολογισμό της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε να συνεχίζει να υφίσταται το ούρπα. Να μην είναι μόνο δηλαδή εξ ολοκλήρου ει βάρο, α πούμε, ή να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να βρούμε μια λύση για το πώς θα χρηματοδοτηθεί μετά την απόσυρση των Αμερικανών. Και τέλο έχουμε και την διάσκεψη δωρητών για την Συρία που θα γίνει στι Βρυξέλλες αύριο και μεθαύριο. Και από αυτό θα υπάρξουν συνέπειες. Πέρα από το 1 δις 275 εκατομμύρια ευρώ από τον κοινωνικό προπολογισμό, Φαντάζομαι ότι θα επιβεβαιωθούν άλλα 560 εκατομμύρια για την περίοδο 2018-2020 και αυτά θα προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη Συρία. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνουν άλλες μετακινήσεις ή περικοπές των κονδυλίων είτε σε σχέση με το εργαλείο για τους πρόσφυγες στην ε, Τουρκία, είτε για το εργαλείο που χρηματοδοτεί την άμυνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε, κύριε Βιώτη, για τις ε, εισηγητικές σας αυτές τις παρατηρήσεις. Όπως είπε ο συνάδελφος, περιμένει να ακούσει τις δικές μας απόψεις. Οπότε θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπενιφέη, μετά στον κύριο Τάνοκ, ο κύριος Καστάλτο έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Μπένιφεϊ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή τη ε, Επιτροπή μα Προπολίου, τον κύριο Βιώτη, που ήρθε εδώ σήμερα, για να συζητήσουμε τι προτεραιότητε για το προεβασμό του 19. Το διεθνέ πλαίσιο εξελίσσεται και θέτει την Ένωση ενώπιον διαφόρων προκλήσεων σύγκρουση στη Συρία έχει μπει σε μια κέρια φάση. Έχουμε τα θέματα που αφορούν το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Έχουμε την κατάσταση στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, ιδιαίτερα μετά την ε, Αραβική Άνοιξη. Υπάρχει η έλλειψη σταθερότητα στην Λιβύη, έχουμε θέματα τρομοκρατίας, έχουμε θέματα διαχείρισης της μεταναστευτικής δροής και απάνθρωπων μεταχειρήσεων. Οι χώρες του Μαστράκη επίσης ε, βλέπουν κάποιες ε, μεταναστευτικές δροές που αποσταθεροποιούν εσωτερικά στις χώρε αυτές. Η Τουρκία πηγαίνει όλο και περισσότερο προς ένα αυταρχικό καθεστώς. Στα Δικά Βαλκάνια έχουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε και την κρίση στην Ουκρανία, η οποία απέχει πολύ από τον αληθή. Αυτά είναι τα πιο κοντινά σενάρια στις πόρτες μας, σε εμάς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ακόμα περισσότερο μια ενεργό και σταθερή εξωτερική πολιτική. Όλοι ε, κάνουν έκκληση για έναν ενεργό ρόλο της Ευρώπης ως παγκοσμίου παράγοντα, ιδιαίτερα τη στιγμή που η Αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει άλλους στόχους και η Ρωσία έχει δική της πολιτική υπερδύναμης αντίθετη με τις δικές μας αξίες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και θα αναφερθώ σε κάποια κύρια σημεία όπως ανέφερε και αυτά προηγουμένως, όπως και αυτά που ανέφερε συγγνώμη προηγουμένως ο κύριος ε, Βιώτη. Οι προτεραιότητες μας παραμένει η εδραίωση της δημοκρατίας, η τήρηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιδών δικαιωμάτων και η προώθηση του κράτους δικαίου και η σταθερότητα κυρίως στις χώρες της γειτονιάς μας. Καταπολέμηση διεθνούς τρομοκρατίας, μείωση της φτώχειας η ανάγκη αντιμετώπισης των αιτιών που βρίσκονται στη ρίζα του ασύλου και των μεταφερικών ροών. Για τα Βαλκάνια η Ιωνία δεν είναι και τόσο θετική, γιατί μετά από την διεύρυνση, το πακέτο διεύρυνσης 18, η στρατηγική του Φλεβάρη προτείνει κάποιες στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχουν επιτώσει όμως τον προϋπολογισμό διεύρυνση των επενδύσεων, ε, δίκτυα διασύνδεσης και κυρίως διπλασιασμός του Εράσμους ΣΥΝ. Είναι ο σωστός δρόμος γιατί το να επενδύσουμε στους νέους είναι κέριο στην Ευρώπη και για τη γειτονιά μας. Οπότε αναμένουμε να επιδοθεί αυτή η δέσμευση. Βέβαια όλα αυτά θα επιφέρουν απαραίτητε αυξήσει στα κονδύλια που θα αφορούν τα Βαλκάνια μέχρι το 2020 και ενδεχομένω θα μειωθούν τα κονδύλια που αφορούν την ε, Τουρκία για την πρόθεση και δρόση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε όμως η πρόταση αυτή να, η πρόταση αυτή να μετατραπεί και σε κάτι αντίστοιχο ε, κατά τη συζήτηση του προπολογισμού στην Τουρκία ας πούμε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κοινωνία των πολιτών. Ε, η ενίσχυση αυτή τη κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να είναι κάτι το αυτόματο, το αυτονόητο σε αυτά τα εργαλεία ενίσχυση και στηρίξη ώστε να έχουμε μια ενίσχυση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Επίση θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εξωτερικές δράσεις. Αναμένουμε μια ενίσχυση των δράσεων οι οποίε ε, δεν θα αφορούν μόνο το ιπα αλλά θα αφορούν και το εργαλείο για την ε, γειτονία στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια που θα αφορούν περιοχές για την ε, γειτονιά της Ένωσης, ε, όχι μόνο Βορεια Αφρική, αλλά Ουκρανία, Γεωργία κλπ. Ενίσχυση επίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι όλο και πιο απαραίτητο λόγω τη τωρινή τάση μείωση ή υποχώρηση τη κοινωνία των πολιτών και τη απειλή που δέχονται τα θεμελιώδη δικαιωμάτων σε πολλέ χώρε. Θα πρέπει εδώ να ενισχύσουμε την, ε, το κομμάτι που αφορά την αποστολή διεθνών παρατηρητών για το εργαλείο τώρα για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Το δεύτερο σκέλος των τριών δις εγκρίθηκε από την Κομισιόν και αυτό παραμένει ένα στατικό στοιχείο επένδυση για την Ένωση. Όμως αυτά θα πρέπει να προέρχονται από διάφορα εργαλεία, όπως το είπα δύο, όπως είπα προηγουμένως, που αφορά την γειτονία. Τώρα, το εργαλείο για τους πρόσφυγες υποβάλλεται και αυτό στι ίδιε διαδικασίε και κυρίω στον λόγο του Κοινοβουλίου. Οπότε βλέπουμε θετικά την πρώτα τροποποίηση του χρηματοοικονομικού κανονισμού που αφορά αυτό το εργαλείο. Αύριο θα ξεκινήσει η διάσκεψη των Βρυξελών για τη Συρία. Οπότε θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε τι δεσμεύσει μα για, ε, για την ανθρωπιστική παρέμβαση και να μιλήσουμε για την ε, νοικοδόμηση. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίω και τα αποτελέσματα και τι επιπτώσει που θα έχουν αυτά στον προπολογισμό του 19. Έχουμε και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θέλει να περιορίσει την δέσμευσή του. Οπότε θα πρέπει εμείς αντίστοιχα να ενισχύσουμε τη δική μας συμβολή. Όπως ακριβώς ε, αναφέραμε στη διασκέψη της Ρώμης, 15 Μαρτίου. Το μακροοικονομικό πλαίσιο για την Ένωση έχει βελτιωθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερα κονδύλια τα οποία θα προωθηθούν ή θα προοριστούν για εργαλεία εξωτερικής ε, δράσης. Πάντως, καταλήγοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κόσμος χρειάζεται μια πιο παρούσα Ευρώπη και δεν μπορούμε παρά να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτή με τα κατάλληλα κοντήλια τις κατάλληλους πόρους για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όπως ε, προσπάθησα να καταδείξω, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις γειτονία μας με τα διάφορα μέτωπα τα οποία υπάρχουν και πάνω στα οποία βεβαίω θα επικεντρωθεί η δουλειά μα, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, thank you to our rapporteur here. Ευχαριστούμε για τον εισηγητή τη Επιτροπή μα, τον κύριο Μπενιφέη. Ε, κύριο Λεωμαρή, έχει το λόγο ο κύριο Γκάλα. Γκάλερ. Κανεί άλλο. Μόνο ΕΛΚ λοιπόν στους ομιλητές. Πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι τις και μισή. Οπότε δύο-τρία λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Κυρία Λιωμαρή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω τις εξής παρατηρήσεις ο προπολογισμό είναι το μοναδικό κριτήριο της ε, πραγματικής, η λιδία λίθο δηλαδή της πραγματικής αποφασιστικότητα για άσκηση πολιτική. Θα ήθελα κύριε Σιγητά να σα ρωτήσω το εξή. Το γεγονός ότι ή ε, βάζουμε, θέλετε να μπουν σε δεύτερο πλάνο ε, τα της αμήνης, ε, μου φαίνεται ότι ε, θα ήταν λανθασμένο. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες θέλουν από εμάς να τους προστατέψουμε. Τα ζητήματα ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας. Η χρημα... Αν η χρηματοδότηση της άμυνας γίνεται μόνο από ό,τι περισσεύει από τα υπόλοιπα κονδύλια, δεν δείχνει ευρωπαϊκή βούληση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους ε, ε, μετανάστες από την Τουρκία. Ε, αυτοί έρχονται κυρίως από τη Συρία. Τελευταία βλέπουμε Σύριους να γυρνούν στην πατρίδα τους. Αντίθετα υπάρχουν άλλοι πρόσφυγες που έρχονται από άλλες περιοχές. Αιθιοπία και άλλες χώρες Αφρικής κυρίως. Εθνικότητες από τις οποίες φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερα προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα επιλογής, πολιτικής επιλογής και δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιοριστούμε να λέμε ότι η προτεραιότητα είναι οι πρόσφυγες από την Τουρκία, ιδιαίτερα σήμερα. Τρίτον, η ε, βοήθεια στην σχέση γειτονία προς την Ανατολή είναι σωστή, αλλά μην αγνοούμε την ανάγκη να αυξήσουμε τη βοήθειά μας στις αφρικανικές χώρες αν θέλουμε να αποφύγουμε μεταναστευτικές ροές εξαιτία δημογραφικών παραγόντων, ε, αστάθειας, λαθρεμπορίου κλπ. κλπ. Τέλος, το να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντισταθμίσει την μείωση των, της ενίσχυσης των ΗΠΑ προς τους Παλαιστινίους δείχνει ότι γινόμαστε σκυλάκι των ΗΠΑ, σαν να εξαρτώμαστε από αυτού και να του συμπληρώνουμε μόνο στην πολιτική του Ευχαριστώ. Next. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δύο λεπτά. Μπορεί και να μην χρειαστώ. Καν δύο λεπτά. Ένα πολύ συγκεκριμένο και σύντομο ερώτημα θέλω να θέσω. Κύριε Πρόεδρε, δε... κύριε Πρόεδρε επαναλαμβάνω, δεν χρειάζομαι δύο λεπτά. Ένα ερώτημα πολύ απλό θέλω να θέσω. Καθώς μιλάμε, με ακούτε. Ωραία. Καθώς μιλάμε, υπάρχουν περίπου σχεδόν 200.000 άνθρωποι που έχουν ε, εκδιωχθεί από το Αφρίν και βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Οι ανάγκες τους είναι πιεστικές και άμεσες και έχω την απορία τι, τι κάνουμε και τι λέμε ε, σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεδομένου ότι συζητούμε και, και μιλούμε τόσο πολύ για τους ε, πρόσφυγες συγκεκριμένο ερώτημα. Μπορούμε να κατανείμουμε τμήμα των τριών δισεκατομμυρίων που έχουμε υποσχεθεί στην Τουρκία. Μπορούμε να πάρουμε ένα τμήμα αυτών, ένα δισεκατομμύριο για παράδειγμα, και να το παράσχουμε στις κουρδικές τοπικές αρχές προκειμένου αυτές να μπορέσουν να καλύψουν κάποιες από τις ανάγκες των προσφύγων που έχουν εκδιωχθεί από την Αφρίν από τα τουρκικά στρατόπεδα. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό χρειαστήκατε τελικά. Κύριε Γκάλερ, είχατε και γενέθλια χθε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. 19 χρόνια συμπληρώνω σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εκτό από τα χθεσινά μου γενέθλια. Έχω να κάνω μια παρατήρηση στον εισηγητή και θέλω να συμφωνήσω με αυτό που είπε η συνάδελφος Αγιομαρή σχετικά με τον τομέα ασφάλειας και άμυνας. Πράγματι, οι προσπάθειες δεν μπορούν ε, να χρηματοδοτηθούν από τα περιθώρια. Έχουμε ευρύτατη ε, συνένεση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, ώστε να ενεργοποιηθεί η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ. Αν δείτε μάλιστα τη συνθήκη, αναφέρει ρητός ότι τα διοικητικά έξοδα, οι διοικητικέ δαπάνες και οι επιχειρησιακές δαπάνες της, της ΠΕΣΚΟ, εφόσον δεν πρόκειται για στρατιωτικές επιχειρήσεις, ε, καλύπτονται από τον ενωσιακό προπολογισμό. Άλλωστε και η Κομισιόν έχει υποβάλει σχετικές προτάσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι καλούμαστε εμείς να θέσουμε μια πολιτική προτεραιότητα η οποία θα αφορά και τον προϋπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δημοσιονομικές προοπτικές ευρύτερα. Και αυτό όχι γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα λεφτά που έχουμε, αλλά ακριβώς γιατί η κατάσταση στον κόσμο έχει πάρει την τροπή την οποία έχει πάρει και ελπίζω αυτή η πολιτική ματιά ε, να, στον προϋπολογισμό να αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ντεγκράντες, τελευταίος ομιλητής. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή, αλλά σας παρακαλώ όσο πιο σύντομα γίνεται. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Μια και είναι εδώ ο κ. Βιώτη, θέλω να πω τα εξή. Ω υπεύθυνο για τι λατινοαμερικανικέ σχέσει στην ομάδα μα, έχω υποβάλει ε, ένα σχέδιο, πιλωτικό σχέδιο για την ε, στήριξη της Κολομβίας ε, μετά την λήξη της, της εσωτερικής σύγκρουσης εκεί. Υπάρχει ένα ταμείο το οποίο βοηθά την Κολομβία, αλλά δεν είναι αρκετή. Το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της Κολομβίας μέχρι το 2030 ε, και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για, τους, για τις ζώνες που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση. Ε, η ΦΑΡΚ έχει δολοφονήσει πολλούς ανθρώπους ε, και πρέπει να τους βοηθήσουμε να είμαστε παρόντες σε αυτή την περιοχή, στην ανοικοδόμηση της ειρήνης με βιώσιμα σχέδια ε, προσθέτοντας στις κρατικές ενισχύσεις και την διεθνή βοήθεια. Η συνεργασία πρέπει να γίνει μέσω τεχνικής συνδρομής και ανάπτυξης ε, ικανοτήτων και προσόντων. Δεν είναι τεράστια τα ποσά, αλλά πιστεύω ότι εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να το δούμε με ρεαλισμό και να συμπεριλάβουμε αυτό το πιλωτικό σχέδιο στον προϋπολογισμό, στις προτάσεις με τον προϋπολογισμό. Παρακαλώ πολύ κύριε Βιώτη, συμπεριλάβετε το ως πολιτική προτεραιότητα. Okay, thank you. No further comments from Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Κύριε Βιώτη, έχετε το λόγο. Μερικά λεπτά για να τελειώσουμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς που μίλησαν που μίλησαν κέρια. Και θα μιλήσω για αυτά που έθιξαν και για αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπενιφέη. Πάντως, να ξεκαθαρίσω το εξή. Δεν θεωρώ, δευτερεύον το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας, έτσι. Ξεκινάμε αυτό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ δεν θέλω να χρηματοδοτηθεί το σκέλος της ασφάλειας και της άμυνας από τα υπολείμματα. Αλλά αν θέλουμε ως χώρες μέλη να χρηματοδοτήσουμε νέα στοιχεία, τότε θα πρέπει να υπάρξουν νέα κονδύλια. Αν λοιπόν οι χώρες μέλη ζητήσουν νέες δεσμεύσεις και νέα προγράμματα, νέα σχέδια, τότε θα πρέπει οι χώρες να συμμετάσχουν, να συμβάλλουν περισσότερο στον κοινοτικό προπολογισμό. Αλλιώ θα υποχρεωθούμε να κάνουμε περικοπέ. Και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε από την λίγα ε, ξύγκη, όπω λέμε, από τον προπολογισμό. Αλλά ξαναλέω, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θεωρώ δευτερεύον το θέμα αυτό. Επίσης να πω ότι συμφωνώ και αυτό που υπόθηκε για το θέμα των Κούρδων για την χρήση των τριών δισεκατομμυρίων όχι μόνο δηλαδή για τους πρόσφυγες, του Σύριου. Και αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε κάθε φορά τα χρήματα αυτά να δοθούν στην κοινωνία των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των κουρδικών αντιστοίχων. Ίσως λοιπόν αυτό σημαίνει ότι Όπως είπε ο κύριος Μπενιφέη, θα πρέπει να έχουμε εργαλεία για να καταπολεμήσουμε τα αίτια και τις ρίζες της μετανάστευσης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίως να βοηθήσουμε και τους πρόσφυγες που υπάρχουν σήμερα. Εγώ είμαι Ιταλός, οπότε ξέρω ακριβώς τι γίνεται και τι ανάγκες υπάρχουν. Και ευχαριστώ για μια φορά τον Πρόεδρο και ευχαριστώ την Επιτροπή σας για τη φιλοξενία και αναμένω την δική σας συμβολή για να δώσουμε τις μάχες εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ. Well, thank you, dear colleague, for your... Ευχαριστούμε συνάδελφοι για τα λόγια σας. Ευχαριστούμε που ε, ήσασταν εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Προθέσεων. Καλή επιτυχία στο σημαντικό σας έργο. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Και περνάμε στο επόμενο θέμα.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 Κυρίε και κύριοι, περνάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 10. Έχουμε την τιμή να καλωσορίζουμε εδώ τον Επίτροπο Γιωχάνες Χάν, που είναι τακτικός προσκεκλημένος μας εδώ στην ΑΦΕΤ και θα μας παρουσιάσει τις εκθέσεις διεύρυνσης που ε, ενέκρινε η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θέλω να ε, συζητήσουμε τόσο συνέχισαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο χαιρόμαστε πολύ που ο Επίτροπος είναι εδώ σήμερα. Και προσκαλέσαμε τον κύριο Χάν να έρθει το συντομότερο δυνατό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα καταφέρατε να έρθετε σήμερα, Δευτέρα. Έχουμε μια πολύ θετική παράδοση να συζητούμε εδώ στην Επιτροπή τις εκθέσεις διεύρυνσης σε βάθος με τον Επίτροπο και θα πρότεινα χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Χάν, που ε, βρισκόταν, αν έχω ενημερθεί σωστά, στα Δυτικά Βαλκάνια, με την ύπατη εκπρόσωπο, τουλάχιστον σε κάποιες από τις χώρες αυτές, και συζήτησε τις εμπειρίες του και τις ε, απόψεις του στις χώρες αυτές, για τις οποίες και θα μας ενημερώσει. Θα πρότεινα λοιπόν να δώσουμε στον κύριο Χάν 10 λεπτά περίπου, ώστε να έχουμε επαρκή χρόνο για απαντήσεις. Ιωάννης Χάν, έχετε παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ. Πράγματι, η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ιδανική όσον αφορά τον χρονικό σχεδιασμό των συναντήσεων και των συνεδριάσεων. Ήταν ένα μείγμα, θα έλεγα, διαφόρων εκδηλώσεων και συμβάντων που δεν μου επέτρεψαν τελικά να παρευρεθώ στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Αλλά ξέρετε ότι προσπαθώ πάντοτε να είμαι διαθέσιμος και στις διμερείς, σας, ε, στις διμερείς επαφές και στις συναντήσεις των πολιτικών ομάδων. Ε, ελπίζω λοιπόν την επόμενη φορά και είμαι βέβαιος δηλαδή ότι θα αποφύγουμε ε, την επανάληψη ενό τέτοιου φαινομένου. Ξέρετε ότι η ομιλία μου αυτή δεν έρχεται μία φορά το χρόνο. Ε, ε, ίσως την επόμενη φορά, ε, θα, μάλλον είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Δεδομένων όλων αυτών λοιπόν, και αφού τα είπα, θα ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω για το πακέτο το οποίο Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από σας έχετε διαβάσει. Βλέποντας και εδώ στην αίθουσα θα ήθελα να καλωσορίσω κάποιους πρέσβεις ε, στην ε, σημερινή μας εκδήλωση. Χαίρομαι που είμαι εδώ, που είμαστε εδώ όλοι. Θα μιλήσω λοιπόν για το πακέτο που εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι ήμουν στα ε, Σκόπια αλλά δεν ήμουνα σε όλες τις χώρες μαζί με την κυρία Μογκερίνη. Εκείνη συνέχισε σε όλες τις χώρες γιατί εγώ ε, μετέβην στην Ουάσιγκτον ε, προκειμένου να συντονίσω τις δράσεις μας με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ιδρύματα ε, και τον Οργανισμό Αραβικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων είναι σημαντικό αυτό γιατί αφορά και τις δικές μας χώρες και τα δικά μας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το πακέτο λοιπόν κάνει ένα απολογισμό της κατάστασης της χώρες και τις, τα συμπεράσματα της ε, εφαρμογής της πολιτικής διεύρυνσης έως και τον Ιανουάριο του 2018 που ήταν η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ε, καθώς αφορά μεταρρυθμίσεις σε θεμελιώδεις τομείς όπως είναι το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, διακυβέρνηση, οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Η Κομισιόν επίσης δημοσιεύει την ετήσια αξιολόγησή της των ε, οικονομικών προγραμμάτων, ε, των ετήσιων οικονομικών προγραμμάτων για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και γι' αυτό συγχρονίσαμε αυτά τα, ε, αυτές τις εκθέσεις, την έκδοσή τους δηλαδή, τη δημοσίευσή τους, τα κάνουμε ε, και για τις δύο περιπτώσεις ε, τον, την Άνοιξη στο πλαίσιο της αξιολόγηση αυτών των ε, προγραμμάτων οικονομικής μεταρρύθμισης. Προφανώς η έκθεση αυτή δεν αποτελεί το τέλος, αλλά μια στρατηγική για την εξαγωγή των δικών μας προτεραιοτήτων στη γειτονία μας. Το πακέτο που παρουσιάσαμε το Φεβρουάριο επανεπιβεβαίωσε για τα Δυτικά Βαλκάνια την ευρωπαϊκή προοπτική της περιφέρειας αυτή και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ε, η έκθεση αυτή αποτελεί έναν απολογισμό αν θέλετε και αποδεικνύει ότι η πολιτική διεύρυνσή μας αποφέρει καρπούς και χαίρομαι πολύ που η Κομισιόν αναγνωρίζει την ηλική και πραγματική πρόοδο που έχουν σημειώσει η Φύρομ και η Αλβανία και ε, συστήνει στο Συμβούλιο να ανοίξει τις ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις και με τις δύο κάνοντα ταυτόχρονα συγκεκριμένε διαπιστώσει ω προ τι ανάγκε να σημειωθεί και περαιτέρω πρόοδο. Και αυτό ε, θεωρώ ότι είναι δείγμα μια ε, πολύ ρεαλιστική αξιολόγηση. Η Αλβανία έχει κάνει μεταρρυθμίσει στη δικαιοσύνη και σε άλλου τομεί, ενώ η ΦΥΡΟΜ έχει υπερβεί μια βαθιά πολιτική κρίση και σημειώνει πρόοδο ως προς τις μεταρρυθμίσεις ε, και τις γειτονικές της σχέσεις. Βεβαίως δεν υπάρχει ε, χρόνος για ε, εφησυχασμό. Ε, οι χώρες λοιπόν έχουν ε, ε, ένα, ε, ένα κοινό, μια κοινή βάση που τις στηρίζει ως προς την ευρωπαϊκή τους πορεία. Βεβαίως η πορεία αυτή θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα σημειωθεί σε επιμέρους τομείς και ε, ένα πράγμα δεν τίθεται ε, υποδιαπραγμάτευση, η ποιότητα έχει προτεραιότητα έναντι της ταχύτητας. Η διεύρυνση λοιπόν δεν αποτελεί χάρη, ε, αποτελεί ζωτικό συμφέρον της ίδιας της Ένωσης και αφορά την δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταίροι μας στα Δυτικά Βαλκάνια γνωρίζουν ότι η διεύρυνση θα γίνει μόνο ε, εφόσον αποτελεί αμοιβαία αποφελή ε, κατεύθυνση. Γι' αυτό και η έκθεση σημειώνει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές. Πολλά πρέπει να γίνουν, ιδίω στους ζωτικούς τομείς του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Στα οικονομικά οι χώρες πρέπει να, υπο να βελτιώσουν το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα και να αντιμετωπίσουν την υψηλή ανεργία και ιδίως την ανεργία των νέων. Να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να προωθήσουν την ατζέντα της συνδεσιμότητας. Η φετινή, ο φετινός λοιπόν συγχρονισμός του πακέτου εκθέσεων με την αξιολόγηση της Κομισιόν για τα ε, προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης της Κομισιόν θα μας δώσουν την δυνατότητα να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα και μια καλύτερη κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν και οικονομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Και τέλος, όλες οι χώρες πρέπει να καταβάλουν ακόμα μεγαλύτερες ε, προσπάθειες στον τομέα της συμφιλίωσης και των καλών γειτονικών σχέσεων. Τα τελευταία, ε, ε τους τελευταίους μήνες είπαμε ότι όλα τα ανοιχτά διμερεί ζητήματα πρέπει να επιληθούν πριν από την ένταξη και ε, το γεγονός ότι το αναφέρουμε αυτό και ρητός ε, στην στρατηγική μας ε, νομίζω ότι άπτεται και οφείλεται μάλλον και στο και στο ότι ήδη κάποιες διμερείς συμ, και διαφορές έχουν ήδη επίλθει. Με τη στρατηγική που παρουσιάσαμε το Φεβρουάριο λοιπόν έχουμε σκιαγραφίσει ε, μια μακρόπνοη στρατηγική για την Ένωση και έχουμε με μεγάλη λεπτομέρεια υποδείξει στις χώρες τι πρέπει να κάνουν. Τώρα πλέον το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των ηγετών των χωρών αυτών για να κάνουν τις δικές τους ε, ενέργειες. Δυστυχώς για την Τουρκία η ανάλυση μας δείχνει ότι η χώρα αυτή εξακολουθεί να απομακρύνεται σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στο τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα έχει καλέσει την Τουρκία να αναιρέσει αυτή την αρνητική ε, πορεία και έχει υποβάλει στην έκθεση συγκεκριμένε συστάσεις προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Ταυτόχρονα η Τουρκία παραμένει στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνω ε, για άλλη μια φορά ε, τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει η Τουρκία προκειμένου να ε, προσφέρει ε, κατάλημα σε πάνω από 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκτιμά ιδιαίτερο την προσπάθεια αυτή. Το πακέτο διεύρυνση δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο μα έχει τελειώσει. Το επόμενο μεγάλο ερώς, ε, ορόσημο είναι η συνδιάσκεψη που θα γίνει στη Σόφια στι 7 Μαου για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και να περάσουμε το μήνυμα αυτό και στις πολίτες της χώρας. Θα είναι μια συνδιάσκεψη η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς Τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Δυτικά Βαλκάνια, στι μεταφορέ στην ενέργεια και ε, στι τηλεπικοινωνίες. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε πραγματικά ωφέλη καθημερινά τόσο στου ε, πολίτε των χωρών αυτών και στου πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεχιζόμενη ε, υποστήριξή σα προ την πολιτική διεύρυνση και, τον, και τις σχετικές διαπραγματεύσεις και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε πλέον να περάσουμε ε, και στην ε, συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννης, ε, που τήρησες το χρονικό σου όριο των 10 λεπτών. Θα περάσουμε στην ανταλλαγή απόψεων. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Μου έχουν πει ποιος επιτρέπεται να μιλήσει, πότε και για πόση ώρα για να το καταλάβετε πρέπει να γνωρίζετε μαθηματικά. Οπότε μην, μην προσπαθήσετε καν να μου αλλάξετε τη σειρά και τον κατάλογο. Ο κ. Κούκαν έχει στη διάθεσή του 3,5 λεπτά και μιλάει πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπέ, συνάλφη, Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπατε στην αρχή, αλλά θέλω να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Πρόεδρος το σημαντικό είναι αυτό να μην ξανασυμβεί. Ε, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ψηλά στην ατζέντα μας ε, τον τελευταίο καιρό και είναι θετική η εξέλιξη που ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Γιούνκερ το Σεπτέμβρη, συνεχίστηκε με την παρουσίαση της στρατηγικής στο Φλεβάρι και τώρα συνε, ε, ε, συνεχίζεται μέσω των προτεραιοτήτων της Βουλγαρικής Προεδρίας. Χρειάζεται να συνεχίσουμε σε, αυτό το, σε αυτή την οδό ε, και με περισσότερη προσήλωση, με πιο στρατηγικούς τρόπους. Χαίρομαι που οι μεταρρυθμίσεις προοδεύουν στην περιοχή. Και ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει στο ευρωπαϊκό μονοπάτι. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τις συστάσεις για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Μακεδονία, λέει ο Μιλτής, και την Αλβανία. Και οι δύο χώρες έχουν εργαστεί πολύ σκληρά τελευταία για να εξασφαλίσουν αυτή τη σύσταση. Η απόφαση είναι σημαντική και ελπίζω ότι θα επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα και απτά βήματα που πρέπει να κάνουμε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε σαφείς ε, τις ε, ε, προσδοκίες μας. Πρέπει οι μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, να εφαρμοστούν στην πράξη. Αυτό ισχύει και για τον Μαυροβούνιο και για τη Σερβία που ήδη έχουν ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις αλλά και για, τις, και για τις χώρες που προετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη σωστή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις πολιτικές ελευθερίες. Όλες οι χώρες της περιοχής έχουν προβλήματα, κάποια προβλήματα με αυτά τα θέματα. Τέλος, οι χώρες της περιοχής αυτής θα πρέπει να προχωρήσουν στην επίλυση διμερών διαφορών τους. Θέλουμε να δείξουν δέσμευση και προσήλωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τις χώρες για να ξεπεράσουν διάφορες εντάσεις και διαμάχες. Σε ε, αυτή, την έννοια ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν ακόμα περισσότερη ευθύνη. Να τελειώσω λέγοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι δυνατή αν δεν τα διμερεί ζητήματα που εκκρεμούν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πρέντα επίση μου ζήτησε να παρουσιάσω τη δική του άποψη, οπότε μόλι φτάσουμε στη Βοσνία Ριζεγοβίνη θα ξαναζητήσω το λόγο. Ευχαριστώ. I fear so. Uh, thank you. Το φοβάμαι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούκαν. Ο κύριος Πίτσουλα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της ομάδας μας και λυπάμαι που δεν ήταν δυνατόν την περασμένη εβδομάδα να συζητηθούν στην ΑΦΕΤ και να παρουσιαστούν η εκθέση για τη διεύρυνση. Χαίρομαι που σας έχουμε εδώ όμως. Καλωσορίζουμε τις θετικές συστάσεις για τη Μακεδονία, λέει ο Μιλτής, και για την Αλβανία. Η Μακεδονία έχει αποδείξει την γνήσια πολιτική της βούληση. Θα ήταν πολύ σημαντικό όμως η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να συμφωνήσουν μαζί με την κοινωνία των πολιτών για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το φόρουμ για τον διάλογο του Ζαμονέ, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμεύσει. Ορισμένε μεταρρυθμίσει έχουν ξεκινήσει μόλι τώρα, είναι χλιαρέ, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζεται η προσπάθεια. Ε, η... Το Μαυροβούνιο Επίση ε, αξίζει την... Ε, ε Αλβανία επίση ε, αξίζει την σύσταση γιατί έχει προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και εν πάση περιπτώσει το παράδειγμα της θα χρησιμεύσει και σε άλλε χώρε περιοχής. Το Μαυροβούνιο έχει ήδη προχωρήσει αρκετά και αξίζει επένων. Μόλις συμπληρώσει όλους τους όρους ελπίζω ότι θα μπορέσει να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς άλλους όρους. Σε ό,τι αφορά την ε, Σερβία υπάρχουν επικρίσεις στην έκθεση και αυτό επιβεβαιώνει τους φόβους μας. Το κράτος δικαίου παραμένει αδύναμο, ε, ο ρόλος των εξάρτητων αρχών πρέπει να ενισχυθεί κλπ. Ε, το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε, έστω και καθυστερημένα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν καλό βήμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοσυφοπαίδιο, ε, η Κομισιόν χρησιμοποιεί τα ίδια λόγια με πέρσι. Διάλογος με την ε, Σερβία, ε, προ, μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος είναι προτεραιότητες. Επίσης, θα πρέπει να ε, οριστικοποιηθεί η ε, διευθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο. Ε, σε ό,τι φορά την απόψη της κυρίας Κάτι για την Τουρκία, θέλω να πω τα εξής νέο σύνταγμα στην ε, Τουρκία που υιοθετήθηκε από το 51% των ε, πολιτών με αρνητικές όμως εκθέσεις διεθνών παρατηρητών. Το νέο προεδρικό σύστημα δεν εξασφαλίζει τις αρχές δημοκρατίας και πολλά κρατημέλη ζήτησαν από την Κομισιόν να αξιολογήσει τον αντίκτυπο. Στη δική σας έκθεση μαζί με τον κύριο Γιούνκερ και την κυρία Μογκερίνη το υποσχεθήκατε, αλλά ε, στην έκθεση δεν βλέπουμε πολιτικά συμπεράσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμω ήταν σαφές, Αν το καινούριο Σύνταγμα εφαρμοστεί χωρίς θεσμούς που να ελέγχουν και διαδικασίε που να ελέγχουν, θα ανασταλεί διαδικασία ένταξη. Και ε, δεν καταλαβαίνω πως η Κομισιόν εξάγει τα ίδια συμπεράσματα με πριν από ένα χρόνο. Κύριε Πίτσουλα, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στον κύριο Τάνοκ για 3,5 λεπτά γιατί είναι και συντονιστής και εισηγητής για το Μαυροβούνιο. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίζω εκ του ΕΣΥΑ, κύριο Χάν, για το πακέτο αυτό που αφορά 7 υποψηφίες χώρες. Και εγώ ήμουν την περσμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και χαίρομαι που λύθηκαν κάποια ζητήματα και ήρθατε εδώ τώρα να συζητήσουμε αυτό το κέριο ζήτημα σε σχέση με την διεύρυνση. Ιδιαίτερα τη στιγμή που βρίσκομαι στο τελευταίο έτος της θητείας μου για μια χώρα που αποχωρεί. Μετά από το μεγαλύτερο χείρημα ευημερίας και ειρήνης στην Υπηρώ η Μακεδονία, λέει ο μιλητή, έλαβε το πράσινο φω για την έξοδο των διαπραγματεύσεων και ότι γίνονται προσπάθειες για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα που υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία και αντίστοιχα με την Αλβανία υπάρχει μια θετική διέξοδος. Είμαι εισηγητή για το Μαυροβούνιο και χαίρομαι που από αυτού υπήρξε πρόσφατα μία συμφωνία για την οριοθέτηση των συνόρων με το Κασιφοπέδιο και ότι είχαμε και επιτυχείς εκλογές για την Προεδρία του Μαυροβουνίου. Και για το Μαυροβούνιο συγκεκριμένα έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Σχεδόν όλα, περίπου 30 κεφάλαια έχουν ανοίξει και παραμένουν κλειστά προσωρινά τρία. Ήμουν πρόσφατα στην Ποντκόριτσα και η προοπτική του 2025 προκάλεσε κάποιες ανησυχίες που ανέφερε ο κ. Γιούγκερ. Αλλά ε, αποτελεί απλά και μόνο μια ένδειξη και όχι κάτι το δεσμευτικό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση του Μαυροβουνίου. Απλά και μόνο αποτελεί δηλαδή ένα υπολογισμό που αφορά τα επόμενα 5 με 8 χρόνια. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι προτιμότερο να προσχωρούν κατά ομάδε οι χώρε. Βεβαίω υπάρχουν αυτοί που είναι πιο μπροστά, και που είναι πιο πίσω στη δικασία προσχώρηση. Πάντα όμω παραμένουν οι ίδιε οι προτεραιότητε και το λέμε και το ξαναλέμε κάθε χρόνο. Ενίσχυση δηλαδή του κράτου δικαίου, ενίσχυση τη δημοκρατία και των θεσμών τη χρηστή διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι κοινά θέματα. Καταπολέμηση επίση του οργανωμένου κλίματο, τη διαφθορά, ελευθερία των ΜΜΕ, η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων κλπ. Και η Τουρκία βέβαια εδώ παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τον προαλήσαντα. Ακούσαμε προηγουμένως και την παρέμβαση του πρεσβευτή της Κύπρου στην Ένωση σε σχέση με τις παραβιάσεις της ε, Τουρκίας στην Κυπριακή ΟΣ με κάποια προσχήματα το τουρκικό ναυτικό παρεμπόδισε δραστηριότητε άλλη χώρα μέλου, ε, συγκεκριμένα εταιρεία ΕΝΗ, για την ε, έρευνα υδρογόνων αθράκων και άλλα πράγματα κάνει η Τουρκία βέβαια παρόλο που είναι χώρα του ΝΑΤΟ αγοράζει ρωσικούς πυράβλους ε, έκανε την εισβολή στο Αφρίν που οδήγησε στον εκτοπισμό χιλιάδων αμάχων συλλήψεις χιλιάδων γκουλενιστών με προσχήματα. Βέβαια, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, πιστεύω, το δικαίωμα της Τουρκίας να χαρακτηρίζεται ως χώρα υποψήφιος τη στιγμή που έχουμε τα παραβιάσεις. Ευχαριστώ. Εδώ θα σταματήσω πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, άλλοι 20 θέλετε να μιλήσετε, έτσι. Σας παρακαλώ να τηρήσετε τον χρόνο ομιλίας. Ο κ. Μεζωρής για 2,5 λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να το τηρήσω το χρόνο ομιλίας. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Εμείς βεβαίως καλωσορίζουμε αυτές τις νέες εντατικοποιημένες προσπάθειες της Κομισιόν ώστε να γίνει κάτι το πρακτικό και εμπροστοβαρές σε σχέση με τα δικά Βαλκάνια πιστεύουμε ότι η στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια ίσως να το πετύχει. Επίσης καλωσορίζουμε την ορατή και ισχυρή δέσμευση της Βουλγαρικής Προεδρίας και χαιρόμαστε που το Συμβούλιο θα συμφωνήσει για το καθεστώς υποψηφίας χώρας για την Αλβανία και τη Φυρό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πακέτο κατά την απόψη μας. κατανοούμε αυτή την αρχή ρεγκάτα, αλλά βλέπουμε ότι μάλλον ότι δεν θα πρέπει κανείς να μένει πίσω όσον αφορά την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορεί τέλος πάντων να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Επίσης, να ζητήσω από τους αδέλφους να μου πούνε από διάφορες πολιτικές ομάδες, όταν θα έχουμε του χρόνου ευρωεκλογές αν οι κορυφαίοι υποψήφοι, οι Spitzenkandidaten, δεν θα χρησιμοποιήσουν θέματα ιστορικής πολιτικής στις ομιλίες τους για θέματα διεθνούς πολιτικής, ίσως αυτό να ήταν καλό να βοηθήσει εδώ την Επιτροπή μας. Και να υπογραμμίσω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τις προτεραιότητες που απαριθμίζονται στην έκθεση της Κομισιόν. Δημοκρατική θεσμοί, κράτου δικαίου, κεφάλαια 23 τα οποία είναι σημαντικά νέα κεφάλαια για το Μαυροβούνιο, Αυτά είναι τα σημαντικά. Και θα ήθελα βέβαια να, να ακολουθούμε αυτές τις αρχές και στο εσωτερικό σύνολο, όχι μόνο με τις υποψήφιες χώρες. Τέλος θα ήθελα να αφορθώ στο εξή. Θα θέλαμε να υπάρχει μια νέα προσπάθεια σε ένα τομέα ο οποίος μπενόβγαινε στις προτεραιότητες, δηλαδή το περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική. γιατί η κατάσταση ποικίλει από υποψήφια σε υποψήφια χώρα, οπότε είναι καλό να αναφερθεί και αυτός προτεραιότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μέζεριτς. Για το ερώτημά σας προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του, της κάθε πολιτικής ομάδας. Ε, πάντως γνωρίζω ότι ο Γάλλος Πρόεδρος δεν θα είναι candidate τον Μάιο του 2019. Ο κ. Καστάλντο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λέω ο κύριο Καστάλτο. Καταρχά λυπάμαι για το γεγονό ότι παρουσιάστηκε αυτό το πακέτο στο Κοινοβούλιο μια εβδομάδα μετά την έγκρισή του. Εμεί ω Κοινοβούλιο είμαστε σύμμαχοι τη Κομισιόν σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν αισθανόμαστε πάντοτε ότι μα επιφυλάσσεται η καλύτερη δυνατή μεταχείριση. Πάντω, ο χρονισμό είναι κέριο. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρώπη, για την ίδια τη διεύρυνση. Το σταυροδρόμι είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν χώρε οι οποίε πια δεν είναι τμήμα αυτή τη ευρωπαϊκή πορεία και αυτό θα πρέπει να το καταγράψουμε. Και υπάρχουν άλλε χώρε οι οποίε αντίθετα κάνουν σημαντικότερε προσπάθειε επειδή ακριβώ θέλουν να είναι τμήμα τη ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Αναφέρομαι βεβαίω εδώ, στην πρώτη περίπτωση, στην Τουρκία. Ο κατάλογο είναι αιτιάζων είναι μακροσκελής δεν λέω ότι θα πρέπει να συνεργαστούν, δεν πρέπει να συνεργαστούμε την ε, Άγκυρα, όπως τα θέματα ας πούμε ε, μετανάστευσης λοιπά Όμως θα πρέπει να συνεργαστούμε στα πλαίσια ενός ε, ορθού πλαισίου. Διαφορετικά διατρέχουμε τον κίνδυνο να το υποβαθμίσουμε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας και να το εκφυλίσουμε από τη στιγμή που η Τουρκία δεν παρουσιάζει πια τις ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις να, ώστε να αποτελεί χώρα υποψήφιο. Και οι πρόσφατε εξελίξει το επιβεβαιώνουν αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το Μαυροβούνιο. Μόλι γυρίσαμε από μια αποστολή στην Πολυκόριτσα ω αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και βλέπουμε για άλλη μια φορά μια χώρα που επιβεβαιώνει την ευρωπαϊκή της έφεση και τάση χωρί περιορισμού. Θέλει λοιπόν αυτή η χώρα να αξιολογηθεί σύμφωνα με τι δικέ τη ε, δυνατότητε είναι αυτή η υπόψη πορεία τη. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη ομοιογένεια στη διαδικασία προσχώρηση. Οι χώρε των δικών Βαλκανίων βρίσκονται σε διαφορετικέ θέσει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τι συγκεκριμένε πολιτικέ στην κάθε χώρα. Και χαίρομαι που η Κομισιόν ζητάει ένα διαπραγματεύσεων με τη Μακεδονία Ολομιλητή, όπου πέραν των υπαρχόντων ζητημάτων. Έχουμε θέμα του ονόματο το οποίο φαίνεται να πηγαίνει προ μια λύση και έχουμε και το θέμα τη Αλβανία όπου υπάρχει μια απαραίτητη και χρήσιμη επιτάχυνση. Τα Βαλκάνια είναι Ευρώπη και θα αποτελέσουν κλίμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι στο να ζητήσουμε το σεβασμό στα κεφάλαια 23-24, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό με μια προοπτική αναχώρα. Καλή δουλειά σα εύχομαι πάντως, Επίτροπε. Μπορείτε να βασίζετε στην στήριξη δική μας Επιτροπής. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε κύριε Καστάλτο. Και μετά τους συντονιστές θα δώσω το λόγο στους συζητητές. Θα δώσω το λόγο στον συζητητή μας για την ε, Σερβία, τον κύριο Ντέιβιτ Μακάλιστερ. Δύο λεπτά. Κύριε Ιωάννες Χάν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος θέλω να πω ότι το Σαββατοκύριακο διάβασα τις εκθέσεις και χαίρομαι για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές δείχνουν ότι η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται στα καθορισμένα κριτήρια στη δίκαιη αιρεσιμότητα. Σας ευχαριστώ που τηρείτε τις αρχές αυτές. Συμφωνώ επίσης μαζί σας όσον αφορά την αξιολόγησή σας για τη Σερβία. Το Μαυροβούνιο και η Σερβία βρίσκονται στην ε, ε, ηγετική θέση στην προμετωπίδα της διαδικασίας διεύρυνσης, έχουν ε, επιβάλει και εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που αποφέρουν αποτελέσματα, ωστόσο χρειάζονται ακόμη ε, στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα για τη Σερβία. Οι ενταξιακές δραματεύσεις δεν είναι αυτός αλλά αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας εξυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό και ως πεπισμένος κοινοβουλευτικός θέλω να επιμείνω στην ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος στη Σερβία. Και τέλος χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Προέδρου Βούτσιτς να ξεκινήσει εσωτερικός διάλογος ε, όσον αφορά τις μελλοντικες σχεσεις σχέσεις Βελιγραδίου-Πρίστινας. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό και γνωρίζουμε επίσης όλοι ότι η Σερβία και το Κωσυφοπέδιο πρέπει να ε, εμπλακούν σε, έναν, ε, σε μεγαλύτερο βάθος διάλογο. Και τέλος, εργάζομαι επί της, του πρώτου σχεδίου έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Σερβία. Βρισκόμαστε ακόμα σε διαδικασία συζήτηση με την Γραμματεία για το χρονοδιάγραμμα. Κατά πάσα πιθανότητα η έκθεση ε, και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνουν πριν το καλοκαίρι και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια το φθινόπωρο. Αυτά και έχω τη χαρά να, δω, δώσω το λόγο στην κυρία Σλάιν που είναι η συγκίτρια μας για την Αλβανία. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Επιτροπέ Συνάλφη. Μιλώ εκ μέρους του κ. Φλάκενστάιν που είναι ο πραγματικός ηγητής του Κοινοβουλίου για την Αλβανία. Καλωσορίζουμε ειλικρινά τη ε, σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσει με την Αλβανία, η οποία πραγματικά το αξίζει. Η χώρα ξεκίνησε να εφαρμόζει ένα πλήρες πακέτο μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό τομέα που συμπεριλαμβάνει και μια διαδικασία έγκρισης των δικαστών. Ε, παρόλο που οι μεταρρυθμίσει δεν έχουν ολοκληρωθεί, φαίνονται ήδη θετικέ επιδράσεις που έχει σε άλλα σημεία κλειδί του πακέτου. Η πρόοδος στο πακέτο αυτό θα βοηθήσει να προχωρήσει η χώρα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό η Αλβανία να διατηρήσει αυτή την μεταρρυθμιστική ορμή. Η, μετα, διαδικασία αυτή ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος θα διαρκέσει αρκετό καιρό αλλά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει στηρίζει πάρα πολύ τις ε, ε, ευρωπαϊκές προσδοκίες της Αλβανίας. Μέσα από ένα, μια, τέτοια, μια τέτοια μεταρρύθμιση άλλωστε θα είναι χρήσιμη και για άλλες χώρες της ζώνης αυτής. Η ε, Κομισιόν θα πρέπει να παρακολουθήσει στενά την πρόοδο που γίνεται σε όλες τις ε, ε, προτεραιότητες μεταρρυθμίσεων. Και τώρα μάλιστα είναι σημαντικό να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η μεταρρυθμιστική όρμη. Η ομάδα μου εξακολουθεί να έχει όπως και η Κομισιόν ανησυχίες για την πόλωση που επικρατεί στην χώρα διότι αυτό δυσκολεύει τον ε, έλεγχο της κυβέρνησης, ε, για παράδειγμα μέσω του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά πρέπει για να προκειμένου να προοδεύσει η χώρα να υπάρχει και μια θεμελιώδη συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Επίσης, η χώρα θα πρέπει να αναλάβει να στηρίξει μεταξύ άλλων την διαδικασία του Βαραλίου και άλλες διαδικασίες περιφερειακής ε, συνδρομής πολύ σημαντικό για να γίνουν πραγματικότητα οι προσδοκίες τους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σλάιν που μίλησατε εκ μέρους του κύριου Φλέκεστάιν. Τώρα ο λόγος του κύριο Ζελίμοβιτς που μιλάει εκ μέρους του κύριου Βάγκελ νομίζω. Ο κ. Βάγκελ θα ήθελε να υπογραμμίσει εκ μέρους ομάδας μας ότι στηρίζουμε την σύσταση της Κομισιόν ε, να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις για τις δύο χώρες. Το πράσινο φως ε, θα ενθαρρύνει την Μακεδονία, λέει ο να βρει και αμοιβαία αποδεκτή λύση για το θέμα της ονομασίας με την Ελλάδα. Επίσης ε, θα ενθαρρύνει την μεταρρυθμιστική ατζέντα που έχει τεθεί και αποτελεί το πλαίσιο μιας οποιασδήποτε μελλοντική πρόοδου. Η νέα μακεδονική κυβέρνηση ε, με επιτυχία ηγείται της ε, χώρας, έχουν βελτιωθεί οι εθνοτικές ε, σχέσεις και έχουν βελτιωθεί οι θεσμοί η κυβέρνηση πια είναι πιο ανοιχτή και δεκτική σε συνομιλίες, για συνομιλίες με την αντιπολίτευση και την κοινωνία. Ε, η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος ε, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του εγκλήματος και του οργανωμένου ε, και του, και του του οργανωμένου εγκλήματος ε, και της διαφθοράς. Ε, θα πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ε, οι ελευθερίες του τύπου και να βελτιωθούν σχέσεις με τους γείτονες και η οικονομία της αγοράς. Η Μακεδονία θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί πλήρως ε, στη Μακεδονία θα πρέπει να συνεργαστούν πλήρω η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση προκειμένου να ε, οδηγήσουν τη χώρα σε ένα ευρωπαϊκό και ευρωατλαντικό μέλλον. Ε, θα πρέπει στο πλαίσιο του διαλόγου Ζάμουνε που θα ξεκινήσει το Μάιο να διευκολυνθεί αυτή η εθνική συμφιλίωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο, ο λόγος του κύριο Κούκαν γιατί αντικαθιστά τον κύριο Πρέντα. Είχατε μιλήσει ένα λεπτό περισσότερο προηγουμένως, οπότε έχετε ένα λεπτό λιγότερο τώρα. Κύριε Έχει περάσει αρκετός ε, καιρός από τότε που εγκρίθηκε το τελευταίο πακέτο διεύρυνσης. Σημειώνω λοιπόν ότι η αλλαγή κλίματος ε, αφορά την Ευρώπη. Σήμερα είμαστε πιο ανοιχτοί απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντικό είναι να αποτελούμε ε, σταθερή και αξιόπιστη προοπτική για τις χώρες της περιοχής. Ελπίζω το 2025 να αποτελέσει πραγματικό ορόσημο για τις χώρες αυτές υπό τον όρο ότι με σοβαρότητα θα επιδιώξουν ε, τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ένταξη της Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων η καταπολέμηση, η αποφασιστική καταπολέμηση της ε, διαφοράς που δυστυχώς αποτελεί ακόμα εγγενές χαρακτηριστικό στην περιοχή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Πριν από λίγους μήνες ε, επιβεβαιώθηκε μέσω έκθεσης η επιβράδυνση των σχετικών εξελίξεων και διαδικασιών λόγω πολιτικών διαφωνιών. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ε, ένα σαφές μήνυμα στις πολιτικές ηγεσίες της Βοσνίας ότι πρέπει η διαδικασία αυτή να, ανατραπεί και να αντιστραφεί. Γιατί χρειάζεται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εκλογική χρονιά, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται εν ώψη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, παραμείνουν προτεραιότητα. Επίσης, συμμερίζομαι την αίσθηση ε, κατεπήγοντος που ε, περιλαμβάνει η έκθεση όσον αφορά την ε, αναγκαία μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Ε, ελπίζω ότι με τις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. Αυτά λέει ο κύριος Κρίστιαν Ταμπρέντα που είναι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βοσνία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον κατάλογο των εισηγητών συντονιστών και επικεφαλής αντιπροσωπιών και περνάμε ε, σε όλους ε, τους συναδέλφους που, θέλουν, που είναι μέλη της Επιτροπής μας και θέλουν το λόγο. Ζεύκη, Κανιέτε, Ντέλη, Κόβατσεφ, Φρονζουλίκα, Μαυρίδης και Φρόιτ. Βαλέρο, Μέζεριτς και ο κύριος Χατζηγεωργίου. Μήπως υπάρχει κάποιος που ζήτησε το λόγο και δεν τον ανέφερα. Επικεφαλής αντιπροσωπιών. Συγγνώμη. Όπω είπα και αρχικά, χρειάζεται κανεί να είναι πάρα πολύ καλό στα μαθηματικά για να μπορεί να συντονίζει αυτή τη συζήτηση. Συγγνώμη, ε, έχετε το λόγο ξανά. Υπάρχει κάποιο άλλο που έχει έρθει εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση με διάφορε ιδιότητε. Κύριε Πίτσουλα, Γιωχάννη, μπορεί να μείνει μέχρι τα μεσάνυχτα. Τέλεια. Γιατί δεν κάνουμε το εξή, λοιπόν, λέει ο πρόεδρο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μα μέχρι τι 7. Α προσπαθήσουμε όλοι μα ε, να είμαστε σύντομοι, ώστε να δώσουμε ε, το χρόνο, τον απαραίτητο χρόνο και στον Επίτροπο για να απαντήσει. Να δώσω τώρα το λόγο στου ομιλητέ μα. Ξεκινούμε με την κυρία Ζόφκου. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ένα ερώτημα έχω να σα θέσω που είναι Πολύ σύντομα. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Έπειτα από την πρόσφατη ακρόαση που έγινε στην Αμερικανική Γερουσία όσον αφορά την κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται ενδεχομένως για μια αποτυχία τον ε, σχηματισμού κυβέρνησης στη Βοσνία έπειτα από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Γιατί το ε, αμερικανικό ε, Υπουργείο Εξωτερικών φαίνεται να ε, προετοιμάζεται για μια τέτοια διαδικασία ε, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κογκρέσο την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό και το ερώτημα μου προς εσάς. Πώς προετοιμάζεστε για το ενδεχόμενο αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης στη Βοσνία μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτσουλα με τη δεύτερη ιδιότητά σας αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Θέλω να πω και εγώ κάποια λόγια, γιατί είμαι επικεφαλής των αντιπροσωπιών για τη Βοσνία και το Κόσοβο. Και θέλω να πω κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υποθούν. Μετά από πολλές καθυστερήσεις, υποβλήθηκε το ερωτηματολόγιο από την Βοσνία. Δυστυχώ, με βάση διάφορου δείκτε, η χώρα αυτή βρίσκεται κάτω-κάτω όσον αφορά την πρόοδο ε, στην ευρωπαϊκή τη προοπτική. Η Βοσνία ε, Ερζεγοβίνη βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο στη δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν μόνο κάποια βήματα όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμός προς τους δημοσιογράφους και κατά ε, παραβίαση του δικαιώματος ε, ελεύθερης έκφρασης. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει διακοινοβουλευτική συνεργασία που έχει φέρει ε, το αδιέξοδο στις σχέσεις του Κοινοβουλίου της Βοσνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς η πρόοδος που θα σημειωθεί φέτος είναι πολύ μικρή καθώς ε, είναι και εκλογική χρονιά. Επίσης δεν υπάρχει συμφωνία για τον εκλογικό νόμο έπειτα και από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρα. Δυστυχώς όλες αυτές οι εξελίξεις φαίνεται να απομακρύνουν τη Βοσνία από την ευρωπαϊκή προοπτική της. Ευχαριστώ κύριε Πίτσουλα και περνάμε στον κύριο Μέζεριτ που ε, επίσης θα μιλήσει δεύτερη φορά αλλά με άλλη ιδιότητα. Πράγματι, ε, μιλώ εκ μέρους του εισηγητή για το κοσυφοπαίδιο. Όπως ε, αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεσή της, η πρόοδος για το κοσμοπέδιο ήταν ε, περιορισμένη και με χαμηλή ταχύτητα. Γι' αυτό λόγο η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη ξεκινήσει και να εστιάσει όλη τη την ενέργεια στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην πράξη και όχι μόνο να μένουν στο χαρτί. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί τώρα ανάγκημα και η διαφθορά, αλλά και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για ένα ανεξάρτητο πλήρες λειτουργών δικαστικό σύστημα. Βελτίωση χρειάζεται ε, η στήριξη των εισαγγελέων και των δικαστών με προσωπικό και ανεξαρτησία τους. Ε, ε, αυτή τη στιγμή όμως το δικαστικό σύστημα υφίσταται πολύ πολιτική επιρροή. Ε, θα ήθελα επίσης να μιλήσω για τις προσπάθειες κατάργησης των ειδικών ε, ε, δικαστηρίων, το οποίο ε, είναι μια προσπάθεια αρνητική και θα πρέπει να ανασταλεί. Για τη διατήρηση σταθερότητα στην περιοχή θα πρέπει να διατηρηθεί ο διάλογος το, μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ενεργειακός τομέας συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν έχει γίνει σχεδόν καθόλου πρόοδο στο περιβάλλον. Αυτό το τελευταίο σχόλιο είναι δικό μου σχόλιο. Ελπίζω να μπορέσετε να επηρεάσετε κατά κάποιο τρόπο και τους pitch and στην επόμενη ε, προεκλογική εκστρατεία. Πρόεδρος. Γκούι, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ οι διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την ώρα μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το ονοματολογικό να καταλήξουν ε, γιατί αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν σύνολο. Ερχόμενος τώρα στο θέμα της ε, Τουρκίας Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιλαμβάνονται πλήρως τι ακριβώς τρέχει στη χώρα, αλλά επειδή πολύ ο επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη χώρα αυτή, νομίζω ότι αυτό δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν την ε, ανάλογη πίεση έτσι ώστε να δούμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Παραμένουμε για πάρα πολλά χρόνια σε μια μέση κατάσταση στη σχέση μας με την Τουρκία, σε μια in κατάσταση, όπως έχω πει πολλάκις, που δεν αποδίδει τίποτα. Νομίζω ότι ο κύριος Χάν καλύτερα από όλους μας γνωρίζει, νομίζω ότι είναι ο ένατος του χρόνου σαν Επίτροπος για θέματα διεύρυνσης, ότι στο θέμα Τουρκία ουσιαστικά αποτύχαμε. Ε, όλες οι προσπάθειες, όλα τα report, όλα τα ψηφίσματα ουσιαστικά έχουν πεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων. Ε, πολλές του ζητήματος Τουρκία έχουν αναφερθεί και εμένα μου, κάνει, μου κάνει πλέον και κόπο η, η συχνή επανάληψή τους επειδή δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά θέλω να σας πω μια μικρή λεπτομέρεια που διάβασα μόλις προχτές. Πέραν των 600 παιδιών κάτω των τριών χρόνων είναι στις τουρκικές φυλακές. Μόλις προχτές μπήκε στη φυλακή μία μάνα 28 ετών με το παιδάκι της τριών χρόνων. Πού θα πάμε, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα με το να λέμε απλώς στην Τουρκία ότι ε, είσαι χώρα κλειδί ε, νομίζω ότι πρέπει να πάρθει μια τελική απόφαση. Ή προχωρούμε μαζί τους ή διακόπτουμε. Η μέση κατάσταση δεν βοηθά. Επιτρέψτε μου 30 δευτερόλεπτα μόνο κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν μου είχατε πει πόσο χρόνο έχω. Υπάρχει μια αναφορά στην έκθεση που λέει ότι η Τουρκία στήριξε τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Πιστεύω ότι ακόμα και αν η Επιτροπή νομίζει αυτό το πράγμα, δεν έπρεπε να αγνοήσει, δεν μπορούσε να αγνοήσει ότι τα 43 χρόνια κατοχής έχουν ένα εμπράγματο βάρος πάνω στα γεγονότα και επηρεάζουν και τις εξελίξεις όσον αφορά τη λύση. Ευχαριστώ. Thank you, colleague. We now come to Sandra Ευχαριστώ. Ο κ. Κανιέτε τώρα. Η κ. Σάντρα Κανιέτε, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτό το πακέτο με την πρόταση για Μακεδονία και Αλβανία για την άρξη διαπραγματεύσεων για προσχώρηση. Θα είναι οι πρώτε που ξεκινούν εδώ και πέντε χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για όλε τι χώρε των Βαλκανίων. Ελπίζω τον Ιούνιο το Συμβούλιο να δώσει το πράσινο φω για την πραγματική έναρξη των διαπραγματεύσεων. Και κατά την εμπειρία μου και την άποψή μου αυτή η διαδικασία θα θα αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο αντιμετώπισης διμερών διενέξεων στην περιοχή και καταπολέμηση τη διαφθαράς. Θα οδηγήσει σε πολιτική σταθερότητα και θα προωθήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύω επίσης ότι η πρόοδο που έχουν κάνει αυτές οι υποψήφιες χώρες και οι προτάσει τη Κομισιόν θα αντιμετωπίσουν την προσπάθεια και της Ρωσίας για επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια. Το 2025 έχουμε μια ενδεικτική ημερομηνία ώστε να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει ανεναντών για όλε τι χώρε και να μπορέσουν να προσχωρήσουν στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κανιέτε. Ο κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κύριε Πιτροπέ. έχουμε την ίδια ευκαιρία, μάλλον την καλή ευκαιρία, οι χώρες μας να έχουν εμπειρία για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυτές να έχουν στο μέλλον την Προεδρία. Τώρα η Βουλγαρία, μετά η Αυστρία και μετά η Ρουμανία και αποτελούν και μια μοναδική ευκαιρία στο να έχουμε μια τελική λύση. Και αυτή και η ερώτησή μου προς εσάς, Επίτροπε, τι αναμένετε από τη διάσκεψη κορυφής στην Σόφια και και τι προσδοκάτε από τις διασκέψεις στο Λονδίνο και το Βερολίνο, ώστε πραγματικά για τα ελληνικά Βαλκάνια να ευοδοθεί η προσπάθειά μας. Θα χρειαστεί δημοψήφισμα για τους πολίτες της πρώην, δημοκρατίας ε, της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της πρώην της Μακεδονίας. Αυτό θα είναι, φαίνεται σημαντικό σε σχέση με την ισχύουσα συμμαχία συνασπισμό που κυβερνάει εκεί σε αυτή τη χώρα, ενδεχομένω και για το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώ τι θα γίνει με αυτέ τι διαδικασίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην υπονομευτεί η αξιοπιστία όχι μόνο τη περιοχή αυτή, αλλά και ολόκληρη τη Ένωση για αυτά τα θέματα προσχώρηση. Και μετά για το κοσφοπέδιο και τη σχέση Σερβίας-Κοσφοπεδίου. Μήπως θα μπορέσουν να αποτελέσουν αυτές οι σχέσεις μεταξύ τους ένα υπόδειγμα για τις υπόλοιπες σχέσεις στην, στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, επίλυσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βαλέρο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση για τον κύριο Χάν για την Τουρκία. Δεν είπατε πολλά, αλλά είπατε ότι η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είμαστε ακόμα παρόλα αυτά σημαντική εταίρη. Να ακούσω λοιπόν, αυτή είναι η επίσημη απάντηση της Κομισιόν για τη διαδικασία προσχώρησης. Οι συνομιλίε προσχώρησης έχουν σταματήσει. Τι νομίζει η Κομισιόν, ποια είναι η απόψη της. Και μετά, γιατί είδος εταιρικής σχέσης μιλάμε, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Γιατί στην έκθεση βλέπουμε ότι στους διαφορούς τομείς Αναφέρεται ότι βρισκόμαστε σε πρώιμη φάση, υπάρχει ήπια κάτι τέτοια ανεγράφεται εκεί στην έκθεση. Ότι είναι μετριοπαθή τα, τα επιτεύγματα κλπ. κλπ. Γιατί ας πούμε δεν λέμε ότι φέτος δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος. Οπότε στην επόμενη έκθεση για για την Τουρκία αν υπάρξει τι προσδοκάμε. Ή κόβουμε τελείως τους δεσμούς μας όσον αφορά τις ε, διαδικασίε προσχώρησης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Βαλέρο. Ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον, τον Επίτροπο για τι προσπάθειε που έχει καταβάλει στην περιοχή προκειμένου να προωθήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα. Δύο συγκεκριμένα θέματα ποια είναι η δική σας θέση για την ελληνική θέση. Ακούσαμε κάποια ναι για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι για την ε, ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ελπίζω ότι αυτή δεν είναι η τελευταία σύσταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έναρξη Διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να υπάρξουν εξελίξεις και σε αυτό το τομέα. Και δεύτερον, στην ε, σύνοδο κορυφής που θα γίνει ε, Σουφ, στη Σόφια, χρειαζόμαστε μία ισχυρή πολιτική διακήρυξη, όχι μόνο στον, στους πολίτες της περιοχής, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο που να λέει ότι το μέλλον της περιοχής αυτής ανήκει στην Ευρώπη και όχι αλλού. Ελπίζω να καταλήξουμε λοιπόν σε μια ε, τέτοια δήλωση ε, και αναφέρομαι ιδίως στις πέντε χώρες που δεν αναγνωρίζουν ε, το Κόσοβο να κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε να διαφυλαχθεί η ενότητα του πολιτικού μηνύματος στη Σοφία. Αλλά ακόμη και αν δεν καταστεί δυνατή η υποστήριξη του Κωσόβου, παρόλα αυτά να εκφραστεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Και σας καλώ να το προετοιμάσετε αυτό κύριε Επίτροπο, εσείς και η κυρία Μογκερίνη. Ε, ξέρω ότι οι, κατε... προσπάθειες σας ήδη σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται, αλλά σας ε, καλώ να κάνετε ακόμη περισσότερο. Ο κύριος Μαυρίδης. Um, <clears throat> Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, το σχόλιο μου θα είναι πολύ εύκολο μετά από την τοποθέτηση του συναδέλφου. Συμφωνώ 100% και χαίρομαι πολύ που φαίνεται ότι, ότι τα πράγματα ε, προχωρούν στα Δυτικά Βαλκάνια και το μέλλον των χωρών αυτών είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα σχόλιο από τον κύριο Γιούγκερ ή από την κυρία Μογκερίνη σύμφωνα με το οποίο ότι κάποιες άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Τουρκία ή η Ρωσία, έχουν ήδη διεισδύσει στην περιοχή προσπαθώντας να την θέσουν υπό τη δική τους επιρροή. Το ερώτημά μου είναι, έχουμε καθυστερήσει ίσως ε, ως προς την παρουσία μας σε αυτές τις χώρες και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Όσον αφορά την Τουρκία, ένα πολύ απλό ερώτημα έχω να σας θέσω. Πιστεύετε, Επίτροπε, ότι στην ε, Τουρκία υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και θα αποκαλούσατε μια χώρα όπως η Τουρκία υπό την κυβέρνηση Ερντογάν ως στρατηγικό εταίρο για, τους, για τα 3 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες ενώ οι ίδιοι δημιούργησαν πρόσφατα 200.000 νέους πρόσφυγες στη Συρία. Αναφέρομαι, ξέρετε, στην εισβολή τους στο Αφρίν. Εγώ δεν θα χαρακτήριζα μια τέτοια χώρα ούτε βασικό, ούτε σημαντικό, ούτε στρατηγικό εταίρο. Ξέρω ότι πρέπει να ακολουθεί το, η της διπλωματίας, αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές όπου πρέπει να πει κανείς τέρμα φτάνει ως εδώ. Ευχαριστώ ο κύριος Άντρο Ντέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποδέχομαι με χαρά βεβαίω αυτές τις εκθέσεις, αλλά αναλύοντάς τες θέλω να μου πει και ο Επίτροπος ποια είναι η θέση του για τις ε, δηλώσεις του κυρίου Μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο σε σχέση με τη διεύρυνση. Γιατί από τις απογοητευμένες ε, αντιδράσεις ε, που διαπιστώθηκαν στην περιοχή ε, νομίζω ότι πρόκειται για μια οπισθοδρόμηση στο 2014 αυτό που, έχουμε να, αυτό που έχουμε σήμερα πλέον. Διότι κατά κάποιο τρόπο, ε, το είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, το θέμα αυτό αφορά και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτών των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι η αξιοπιστία αυτή επλήγει πέρσι. Ε, λόγω της στάσης και των δηλώσεων του κυρίου Μακρόν ε, που έγιναν δύο μόλις μήνες μετά την παρουσίαση της στρατηγικής κομισιόν και βλέποντας όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Βουλγαρική Προεδρία αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη που είναι υπέρ της διεύρυνσης και βεβαίως και των δικών, ε, έχοντας υπόψη και τις δικές μας προσπάθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, το να περιμένει κανείς ε, να ολοκληρωθούν ε, οι μεταρρυθμίσεις προτού ενταχθούν αυτές οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μειοπικό γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της σταθερότητας και τις ανάγκες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Θα ήθελα λοιπόν την δική σας θέση επί των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ Άντρο Ντέλη. Σύμφωνα με τον κατάλογό μου, ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Φρόιντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα επανέλθω σε αυτά που είπε ο κ. Φραντζουλικά για τα θετικά αποτελέσματα που μπορούμε να περιμένουμε από τις ε, επόμενες προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα διαφωνήσω ότι αφορά την Αυστρία. Από όσα έχω ακούσει, Οι προτεραιότητες είναι το, η ασφάλεια, το Brexit και η επικουρικότητα για την ε, Προεδρία της ε, Αυστρίας. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Οπότε κύριε Επίτροπε, εσείς, μιλώντας με τον Αυστριακό Πρωθυπουργό, έχετε προσπαθήσει να επηρεάσετε την κυβέρνηση Αυστρίας με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να δώσουν έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια. Δυτικά Βαλκάνια τα οποία ε, λόγω της ε, ιστορίας τους ε, έχουν μια εγκύτητα με την Αυστρία. Πάντοτε η Αυστρία είχε καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες και θα έπρεπε να ενδιαφέρεται. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Ο λόγος του κύριο Χάν Απαντήστε όσες ερωτήσεις μπορείτε. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να τη ομαδοποιήσω. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει την ίδια αξιολόγηση. Δεύτερον, όλοι γνωρίζετε την θέση των κρατών μελών. Τις θέσεις των κρατών μελών. Από όσο γνωρίζω, μόνο μία χώρα είναι σαφώς υπέρ της ε, αναστολής ε, των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Όλες οι άλλες χώρες θέλουν να διατηρήσουν τις πόρτες ανοιχτές. όπως και εσείς μας ζητήσατε βέβαια και αυτές μας ζήτησαν να ε, ξαναδούμε το θέμα της χρηματοδότησης και το κάναμε. Αναθεωρήσαμε τη χρηματοδότηση. Ε, στην ε, ενδιάμεση έκθεσή μας ήμασταν πιο αισιόδοξοι από ότι οι δύο συνομοθέτες. Η πρόταση ήταν 100 εκατομμύρια συν 75 εκατομμύρια για το αποθεματικό. Αυτή ήταν η τελική απόφαση σε συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Οπότε ας μην μπούμε σε μια ε, μάχη, σε ένα αγώνα για το ποιος θα κόψει περισσότερα. Ας δούμε πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία καλύτερα. Η κατάσταση είναι προφανής. ε, οι ενταξιακές διαπραγματεύσει ε, είναι στάσιμες. Εγώ όταν λέω ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός ε, εταίρος κλειδί, ε, νομίζω ότι αναφέρουν πιο πολύ στο μέγεθός της, στον πληθυσμό της, την γεωστρατηγική της σημασία, τις εξωτερικές και εσωτερικές απειλές που δέχεται. Οπότε Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μας ε, σπρώχνουν στο να διατρούμε στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία. Οι ε, υπερχόμενες εκλογές νομίζω ότι προκυρήθηκαν και για οικονομικούς λόγους. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία χειροτερεύει και δεν θα θέλαμε, δεν θα ήταν προς μας να επικρατήσει αστάθεια. Ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά θα θέλαμε μια ανάστατη Τουρκία. Δεν είναι προ συμφέρον μας. Αν το πολιτικό περιβάλλον το ευνοήσει, θα ε- θέλαμε να ζητήσουμε διαπραγματευτική εντολή για την αναβάθμιση της τελωνιακής σχέσης, για παράδειγμα. Θα ήταν προς κοινό συμφέρον και των κρατών και της Τουρκίας μια αναθεωρημένη ε, και αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση. Τώρα, οι επερχόμενες εκλογές και ιδιαίτερως η προεκλογική εκστρατεία στην Τουρκία και ελπίζοντα, ελπίζω όχι εκτός Τουρκίας, δεν, ελπίζω λέω δεν θα συνεισφέρει στην αύξηση των εντάσεων και των παρανοήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ελπίζω ότι η, ο Ερντοάν και η ε, βοηθή του, ε, η συμβουλή θα το καταλάβουν. Ελπίζω οι δύο επόμενοι μήνες της προεκλογικής εκστρατείας να μας βοηθήσουν να μπούμε σε μια πιο λογική σχέση, πιο ανθρώπινη σχέση. Σαφέστατα έχουμε διαφωνίες σε διάφορους τομείς και έχουμε επικρίνει όχι μόνο σε εξελίξεις τις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και παραβιάσεις συνόρων κλπ. Ε, αν δεν ήμασταν απαρκώς σαφείς, θα είμαστε σαφείς στο μέλλον. Αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε και το γεγονός ότι η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες, ε, είναι αξιοσημείωτοι γείτονες και το συμφέρον μας είναι να το ε, κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο πήρε την απόφαση που πήρε. Τώρα για άλλες χώρες. Το θέμα το ονοματολογικό. Ε, είμαι αισιόδοξο ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε μία λύση. Τουλάχιστον μία λύση που θα στρώσει το δρόμο, θα ανοίξει το δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την ΦΥΡΟΜ. Όλοι νομίζω συμφωνούν ότι κάτι θα ήταν χρήσιμο για την χώρα, για την κοινωνία και για όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για την Αλβανία. Κωσυφοπαίδιο. έχουν λάβει χώρα ε, ε, γεγονότα που δεν είναι θετικά. Για παράδειγμα την έκδοση, όπως θέλετε πέστε το, έξι πολιτών στην Τουρκία, χωρίς να τηρηθούν βασικοί κανόνες του κράτους δικαίου. Απ' την άλλη μεριά το Κοινοβούλιο του Κοσμοπεδίου είχε την ευκαιρία να υιοθετήσει τις νομικές διατάξεις ό,τι αφορά το θέμα του καθορισμού των συνόρων. Αυτό είναι θετικό. Ε, έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική. Είχαμε πει ότι δεν θα δεχτούμε στους κόρπους μας οποιοδήποτε νέο μέλος που θα έχει εκρεμής, εκρεμή προβλήματα, ανεπίλητα προβλήματα με τους γειτονές του. Ε, η, ο καθορισμός των συνόρων, αν επιτύχει, δεν θα είναι προς όφελος της Ελβίας, θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Θα έδινε και στις δύο αυτές χώρες μια όθηση. Αυτό νομίζω έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν όλοι σε αυτή την περιοχή. Για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Δεν θέλω να προδικάσω το τι θα γίνει αν οι εκλογές δέλα μου χώρα με τις εγγύσεις τις οποίες θέλουμε να δούμε κλπ. Σίγουρα θέλουμε να είναι ε, σωστές οι εκλογές και το αποτέλεσμα να αναγνωριστεί έτσι ώστε να έχει να φέρει ε, ε, αποτέλεσμα και στη χώρα. Θέλουμε να διευκολύνουμε μια οποιαδήποτε συμφωνία προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά είναι σημαντικό όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι οι πολιτικοί να γνωρίζουν τις ευθύνες τους και να τις αναλάβουν. Αν δούμε τις φημομετρήσεις, μιλώντας με πολίτες της χώρας, ιδιαίτερως νέους, πολίτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ακόμα και όταν δεν είμαστε στη Βοσνία αλλά αλλού στην Ευρώπη, όλοι μας ζητούν, όλοι μου ζητούν να τους υποστηρίξουμε στην ευρωπαϊκή τους προοπτική. Νομίζω ότι υφίσταται ο φόβος μήπως μείνουν πίσω σε σχέση με άλλους στον αγώνα αυτό ένταξης. Ε, στη χώρα υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες, έχουν διαφορετικά ενδεχομένω συμφέροντα, αλλά χρειάζεται η χώρα να κατασκευάσει ένα εθνικό όραμα, να χτίσει ένα εθνικό όνειρο και εμείς είμαστε έτοιμοι να τους διευκολύνουμε, αλλά θα πρέπει εκεί η υπεύθυνοι πολιτικοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εγώ να εμπλακώ ακόμα περισσότερο έστω και προσωπικά αν υπάρχει οποιοδήποτε, ε, οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχουν σκεφτεί κάποια λύση στο μυαλό τους, έστω και στο μυαλό τους. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, Προεδρίας Αυστρίας, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μία από τις κεντρικές προτεραιότητες και το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει. Και ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα με ρώτησε αν μπορούμε να επισκεφθούμε από κοινού την περιοχή, να διοργανώσουμε συνέδρες, συναντήσεις εκεί και η Ρουμανική και η Κροατική Προεδρία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Αλλά προφανώς και άλλες χώρες που δεν είναι, έχουν ακόμα την Προεδρία, όπως η Γερμανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνάντηση της Σόφιας. Όπως κάναμε και με την Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής και της Γειτονίας, ε, εστιάζουμε στο να έχουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα που να στηρίζει τις προσδοκίες, τις ευρωπαϊκές προσδοκίες των χωρών της περιοχής. Ε, καλύτερη συνδεσιμότητα ε, και στην ενέργεια και στο ψηφιακό τομέα, όχι μόνο στις μεταφορές και τα δίκτυα. Ε, η καλύτερη ε, καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Αυτά είναι απαραίτητα, γιατί αν δεν τα κάνουμε, αν δεν προχωρήσουμε εκεί, δεν θα προχωρήσει και η ένταξη, η ευρωπαϊκή πορεία. Είναι πολύ σημαντικό άλλωστε και για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, της περιοχής. Έχουμε πολύ δυναμικό το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αχρησιμοποιητό. η ενίσχυση της οικονομίας πυροδοτεί μεταρρυθμίσεις και στο κράτος δικαίου αμέσως. Ε, προφανώς εκεί έχουμε αδυναμίες, αλλά προτιμάμε να μιλάμε για τα θετικά, γιατί αυτά μπορούν να πυροδοτήσουν, όπως λέω, βελτιώσεις και εκεί που έχουμε αδυναμίες. Θα ζητήσω από τους ε, συνεργάτες μου να εστιάσουν περισσότερο στη λειτουργία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων. Τα ανώτατα δικαστήρια δίνουν κατευθυντές γραμμέ για το πώς θα αξιολογηθούν ορισμένε περιπτώσεις. Αλλά τελικά τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια είναι αυτά τα οποία κάνουν τη δουλειά και που είναι αυτά με τα οποία έρχονται σε επαφή οι πολίτες. Ελάχιστες περιπτώσεις φτάνουν στον το δικαστήριο, οπότε η ποιότητα, η ανεξαρτησία, η διαφάνεια των δικαστηριών φαίνονται ιδιαίτερα στην ποιότητα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων. Αυτό πρέπει να το δούμε για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της, ε, της ενδεχόμενης αποκέντρωσης. Και να εξετάσουμε την απόδοση και την ποιότητα των τοπικών αρχών και κυβερνώντων. Πολλοί επιχειρηματίες εντός και εκτός της περιοχής αυτής μου αναφέρουν και καταγγέλουν περιπτώσεις διαφθοράς και πολύ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Άρα λοιπόν η πρόοδος ε, των χωρών αυτών σχετίζεται με την πρόοδο και σε, σε τοπικό επίπεδο. Σερβία. Κάναμε την αξιολόγησή μας. Η Σερβία είναι παίχτης κλειδί στην ζώνη αυτή. Ε, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και θαραλέα προσπάθεια διαλόγου είναι σημαντικό να αντιδρούμε ψύχρεμα, πιο ψύχρεμα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε τα μάτια σε υπάρχουσες αδυναμίες στο κράτος δικαίου. Έχουμε ένα οδικό χάρτη, τον οποίο έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, την υλοποίησή του. Μέχρι το τέλος του 2016 έπρεπε να είχαμε κάποια μέτρα, που δεν έχουν υιοθετηθεί. Είμαστε στο 18 πλέον και ακόμα δεν τα έχουμε δει. Και οι Σέρβοι πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε όλα τα μέτωπα. Δεν είναι αρκετό να είναι πολύ καλή σε ένα θέμα και όλα τα άλλα να τα περιθωριοποιούν. Και εδώ έρχομαι στο τελευταίο, στην τελευταία παρατήρηση που έχω να κάνω. Για την ομιλία του κυριτού Πρόεδρου Μακρόν και τις αντιδράσεις. Είναι καλό παράδειγμα και απόδειξη της σημασίας της στρατηγικής μας α, αφενός ε, ε, το ότι, ε, το ότι ε, αναφέρθηκε μία μόνο ημερομηνία, το 2025. Τώρα η κατάσταση και εντός και εκτός της ε, περιοχής γίνεται πιο συγκεκριμένη. Μέχρι τώρα ήταν ανέφελο. Ποσχέσεις, ευρωπαϊκή προοπτική, όλα αυτά ήταν λίγο θεωρητικά ή δεν ήταν πολύ, πολύ πραγματικά. Τώρα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία όλα έγιναν πιο απτά. Και μέσα από τι ανησυχίε είναι κατανοητές. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία άσκησε θετική πίεση σε όλες τις πλευρές. Και στην περιοχή για να εργαστούν σκληρά και να πετύχουν. Οι πολίτες πια ξέρουν ότι είναι δυνατόν υπό την προϋπόθεση ότι οι ηγέτες θα είναι υπεύθυνοι, αλλά δραθετικά και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχουν απόλυτα θεμητά κατανοητά επιχειρήματα ε, υπέρ της βελτίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα και να είμαστε προδραστικοί Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν το φθινόπωρο θα υποβάλει πρόταση τομέων όπου πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να περάσει από την ομοφωνία στην πλειοψηφική λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να είμαστε πρώτα δραστικοί όπως λέω να επηρεάζουμε τις διαδικασίες και να αποφασίζουμε πραγματικά ποιο θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα ε, και σε περιφερειακό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια τέτοια εσωτερική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως απαραίτητη. Αλλά πιστεύω ότι και τα δύο πρέπει να γίνουν παράλληλα δεν θα ήταν δυνατόν να περιμένουμε χρόνια μέχρι ότου εμείς συμφωνήσουμε κάτι προκειμένου να συνεχίσουμε μετά με τις ε, διαδικασίες, τις ενταξιακές διαδικασίες. Αντιθέτως, τη χρειαζόμασταν αυτή τη θετική πίεση για να εξετάσουμε πώς θα διορθωθούμε καλύτερα εσωτερικά, ε, πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και σίγουρα υπάρχει πολύ περιθώριο βελτίωσης. Οπότε τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Τέλος, και κατά κάποιο τρόπο συνοψίζοντας, να πω ότι πρέπει να ε, έχουμε στο μυαλό μας ότι αν οι εταίροι μας υλοποιούν τα συμφωνηθέντα, πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Αυτό έχει σχέση με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θεωρούμαστε soft power, με τριοπαθής δύναμη και είμαστε. Το βασική μας αρετή είναι η αξιοπιστία μας ε, και η λογοδοσία μας το ότι δίνουμε λόγο για τις πράξεις μας. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να ξεκινήσετε αυτή τη συζήτηση, αυτό το διάλογο στις χώρες σας γιατί είναι προπετούμενο για μια μελλοντική, οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση. Mm. Πάντως πρέπει αυτά τα δύο να γίνουν παράλληλα. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και η εσωτερική διαβούλευση. Ευχαριστώ πολύ και για το ενδιαφέρον σας και για την στήριξή σας. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είστε πάρα πολύ δραστήριοι στην ΑΒ χώρα. Και θα ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να έχει ε, αντιπροσωπείες, γραφεία σε αυτές τις χώρες. Το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Ε, θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό τις ε, διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί και στο κοινοβουλίο τους και γενικά στο εσωτερικό των χωρών αυτών. Θα, ήταν, θα είχαν να παίξουν αυτές οι αντιπροσωπείς ρόλο κλειδί στην ένταξή τους. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Πριν πεταχτείτε και φύγετε, συναδελφοί, να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο για τα γεγονότα της περσμένης εβδομάδας στο Στρασβούργο. Να πω κάτι ξεκάθαρα. Δεν αποφασίζει ο Επίτροπος Χάν για το χρονοδιάγραμμα του συλλογή των επιτρόπων, το συνεδριάσεων του δηλαδή. Αυτό αποφασίζεται σε άλλη φάση. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν καλή ιδέα να παρουσιάσουμε την έκθεση για διεύρυνση στο Στρασβούργο. Οπότε αν θέλετε μπορώ να γράψω μια επιστολή από τώρα στον πρόεδρο Γιούγκερ ζητώντας να γίνει η επόμενη παρουσίαση του πακέτου διεύρυνσης στις Βρυξέλλες. Γιατί αυτή τη φορά μακρηγόρησε ο κύριος Μακρόν. Πώς να ξέρουμε ποιος θα μιλήσει τον Απριλίου του 2019. γιατί τότε θα έχουμε την επόμενη έκθεση. Οπότε ας προσπαθήσουμε να βρούμε μια ημερομηνία για τις Βρυξέλλες και να το καταστήσουμε σαφές προς τον πρόεδρο της Κομισιόν. Να ευχαριστήσω πάντως τον κύριο Χάν που ήρθε σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Και ας συνεχίσουμε να προσπαθούμε από κοινού ώστε να είναι επιτυχής η διεύρυνση. Σας ευχαριστώ. για τη συνεδρία σας.